Dear colleagues, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε σε ένα λεπτό. Παρακαλώ να καθίσετε στις θέσεις σας. Ja, så går vi i gang. Jeg håber, at I tager høretelefonerne på, fordi jeg har tænkt mig at tale på dansk i dag. Godt. Jamen, velkommen til den her workshop. Λοιπόν, θα ήθελα να σας χαιρετήσω σε αυτό το εργαστήριο, σε το workshop της Επιτροπής για την Ιστορική Αγορά και θέματα των καταναλωτών. Ο σκοπός της σημερινής συνεδρίας συζήτησης είναι να φωτίσουμε το θέμα, το θέμα της οδηγίας για την ασφάλεια των προϊόντων και να δούμε πώς, κατά πώς, να εξοργήσουμε κατά πώς είναι τόσο καλή όσο αναμέναμε. Γιατί αποτέλεσε ακρογωνία ολίθο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να την εξολογήσουμε. Θέλουμε επίσης να ξέρουμε κατά πόσο λειτουργεί εύρυθμα η ιστορική αγορά, κατά πόσο υπάρχουν αδυναμίες ή όχι. Θα πρέπει να αλλάξουμε. Και ο τρίτος τομέας είναι το νέο νομοθετικό πλαίσιο και κατά πόσο μπορεί να συνδυαστεί με την οδηγία για την γενική ασφάλεια των προϊόντων. Θα προσπαθήσουμε να λύσουμε κάποιες, κάποια στοιχεία για την διατύπωση συστάσεων σε σχέση με τα θέματα αυτά από τη σημερινή συζήτηση. Εγώ είμαι η συγγήτρια και θα κάνω μία παρουσίαση ο σκοπός μας είναι να εξασφαλίσουμε για τον καταναλωτή μια ασφαλή προϊόντα. Ε, ήθελα να φέρω μαζί μου αρχικά την βοηθό μου. Er Έχουμε εδώ αυτό το, αυτή την κουρτίνα, το παραπέτασμα το οποίο μπορεί κανείς να το αγοράσει σε διάφορα καταστήματα στην Ολλανδία. Εγώ το έχω σπίτι μου στο παιδικό δωμάτιο, αλλά το πρόβλημα εδώ είναι ότι θα μπορούσε κανείς να στραγγαλιστεί με αυτή την κουρτίνα, την κρεμαστή κουρτίνα. Για παράδειγμα, ένα παιδί θα μπορούσε να πνιγεί με, αυτό το, με αυτή το σκηνή. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει να απολύτει το προϊόν αυτό. Ε, πρόκειται εδώ για ένα κενό στην εποπτεία της αγοράς ή στην ασφάλεια των, γενική ασφάλεια των προϊόντων. Υπάρχουν τέτοιου είδου συγκεκριμένα προϊόντα για παράδειγμα, παιδιά τα οποία πεθαίνουν ακριβώς επειδή στραγγαλίζονται με αυτά τα σκηνιά ή αυτές τις κορδέλες. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει πιο αυστηρή η νομοθεσία σε σχέση με αυτά τα προϊόντα. Ή ένα άλλο παράδειγμα, αυτό εδώ το στυλό, το οποίο το αγόρασα εδώ κάτω στο κοινοβούλιο, στο κατάστημα. Μοιάζει με κραγιόν, αλλά είναι στυλό. Εάν το ανάψει κανείς, ε, υπάρχει εδώ ένα μικρό φως και μπορεί κανείς να το χρησιμοποιήσει για να γράψει. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι, είναι στυλό. Αλλά έχει ένα, μια μορφή που είναι αρκετά ελκυστική για τα παιδιά. Και ανακύπτει λοιπόν το ερώτημα κατά πόσο χρειαζόμαστε ειδικού κανόνε, ειδικά για εκείνα τα προϊόντα που είναι ιδιαίτερα ελκυστικά για τα παιδιά. Γιατί είναι μεν μπορεί κανεί να το χρησιμοποιήσει για να γράψει, αλλά λόγω του χρώματο και του φωτό προσελκύονται παιδιά από αυτό το προϊόν. Και μία μικρή πεντάχρονη πριγκίψα θα ήθελε να παίξει με αυτό το προϊόν, τη πέφτει κάτω, ε, σπάει στη μέση και το καταπίνει. Λοιπόν, αν και το, το ερώτημα κατά πόσο θα πρέπει τα προϊόντα αυτά να συνοδεύονται από, μια, από κάποιες ειδικές διατάξεις, προστασίες για τα παιδιά. Προϊόντα τα οποία είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ελκυστικά για τα παιδιά θα πρέπει να συνοδεύονται ή να πληρούν ειδικέ ε, προδιαγραφέ ασφαλεία. Θα ήθελα εγώ προσωπικά μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Όλοι εδώ έχουμε τον ίδιο σκοπό, τον ίδιο στόχο, θέλουμε μια ασφαλή εσωτερική αγορά για τα προϊόντα μας και ναι μεν έχουμε αρκετές διατάξεις, κανόνες ασφαλείας αλλά επιδέχονται κάποιων βελτιώσεων. Σήμερα έχουμε 7 ομιλητές, δύο ώρες στη διάθεσή μας. Θα πρέπει να τηρήσουμε τα χρονικά μας όρια αλλά χρειαζόμαστε πραγματικά μια πλατιά προοπτική, ιδιαίτερα όσον αφορά την παρακολούθηση, την εποπτεία της αγοράς. Το πρόγραμμά μας γι' αυτό είναι κάπως φορτωμένο. Εγώ θα είμαι αρκετά αυστηρή ως πρόεδρος γιατί θέλουμε να επιτρέψουμε και κάποια ερωτήματα ή σχόλια των βουλευτών. Έχουμε βουλέψει δύο τμήματα στην ακρόασή μας. Καταρχήν, μία μελέτη για την οδηγία για την ασφάλεια των προϊόντων και την επιτήρηση της ε, αγοράς και στη συνέχεια θα ακούσουμε την άποψη της Επιτροπής και ακολούθως έχουμε τη Business Europe και τους δικούς τους εκπροσώπους, πώς βλέπουν εκείνοι τα πράγματα. Και τέλος υπάρχει η δυνατότητα για ερωτήματα και απαντήσεις εκ μέρους του πάνελ. Λοιπόν, Χαίρομαι πάρα πολύ για τις ομιλίες που θα ακολουθήσουν. Η πρώτη ομιλήτρια είναι η Χάνα Μάγια Κούν από τη Rumble Management. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you, Madam Chairwoman. Um, um, Ευχαριστώ πολύ, αγαπητά μέλη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δώσετε την ευκαιρία να έρθω εδώ και να παρουσιάσω αυτή τη σύντομη ομιλία για την αναθεώρηση της ε, οδηγίας για την ασφάλεια των προϊόντων. Θα ήθελα να ξεκινήσω παρουσιάζοντας τους ε, στόχους της ε, μελέτης μας. Καταρχήν, ε, θελήσαμε να αναλύσουμε αυτή την οδηγία για τη γενική ασφάλεια τροφίμων και το νέο νομοθετικό πλαίσιο και να παράσουμε μία εποπτεία ε, ενδεχόμενων αποκλήσεων μεταξύ των δύο. Στη συνέχεια, εξετάσαμε κατά πόσο υπάρχει μία ανάγκη ευθυγράμμισης μεταξύ των δύο και είχαμε κάποιες επιπλέον ερωτήσεις όσον αφορά την παρακολούθηση της αγοράς, την εποπτεία της αγοράς. Καταρχήν θελήσαμε να τονίσουμε τις υπάρξεις εμπειρίες όσον αφορά τις κοινέ δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς και επίσης θελήσαμε να εξετάσουμε την ανάγκη εποπτείας της αγοράς που σχετίζεται ειδικά με τους καταναλωτές για να δούμε κατά πόσο τέλος υπάρχει ε, κατά πόσο είναι ενδεδειγμένη η φυστάμενη νομοθεσία. Ε, σε σχέση με την ασφάλεια προϊόντων. Και θα προσθέσω τώρα τα βασικά συμπεράσματα της έρευνάς μας. Όσον αφορά την εφαρμοσιμότητα της ε, οδηγίας και το νέο νομοθετικό πλαίσιο και την τομεική νομοθεσία. Η οδηγία για την ασφάλεια προϊόντων αφορά όλα τα μη καταναλωτικά προϊόντα, ε, μπορείτε να την ονομάσετε ένα δίκτυο ασφαλείας γιατί αφορά εκείνες τις περιπτώσεις όπου η τομεακή νομοθεσία δεν είναι ειδική. Είναι τμήμα του νέου νομοθετικού πλαισίου και εφαρμόζει κάποια προϊόντα αποκαλύπτονται από την ε, τομεακή νομοθεσία, την εναρμονισμένη νομοθεσία. Και υπάρχουν ορισμένε επικαλύψει μεταξύ των δύο. Όταν, για παράδειγμα, πρόκειται για την εναρμόνιση των καταναλωτικών προϊόντων. Και ο γενικό κανόνα εδώ είναι ότι η, οδηγία, η Γενική Οδηγία για την Ασφάλεια Προϊόντων αφορά πιο ειδικέ περιπτώσεις από το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Τώρα, όσον αφορά την τομαϊκή νομοθεσία, μπορούμε να πούμε ότι η τομαϊκή νομοθεσία έχει μια προτεραιότητα σε σχέση με τις διατάξεις στη νέα οδηγία για την ασφάλεια των προϊόντων ε, και υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που είναι πιο ε, ειδική η τομαϊκή νομοθεσία. Ε, υπάρχει και η απόφαση του 2008 που είναι τμήμα του νέου νομοθετικού πλαισίου και αφορά Κάποιε ε, διατάξεις σχέση, αναφορά σχέση με την εναρμόνιση. Αυτά λοιπόν είναι τα τρία νομοθετικά πλαίσια. Τώρα, όσον αφορά τα συμπεράσματά μα, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν πράγματι κάποιε διαφορές στους ορισμούς μεταξύ του νέου νομοθετικού πλαισίου και την οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων ε, σε σχέση με του ε, οικονομικού φορείς και το πώ τοποθετούνται τα, τον ορισμό και το πώς τοποθετούνται τα προϊόντα στην αγορά. Ωστόσο, οι διαφορές και οι αυτέ αυτές δεν είναι σε επικίνδυνε υπό την έννοια ότι δεν ε, θέτουν σημαντικέ ε, προκλήσει για την ασφάλεια των καταναλωτών και την εποπτεία της αγοράς. Ωστόσο, αυτοί με τους οποίους κάναμε συνεντεύξεις που είναι οι εκπρόσωποι των, ε, από 10 χώρε μέλη και από διάφορες οργανώσει ε, καταναλωτών, καθώς και εκπροσώπους των Γενικών Διευθύνσεων της Επιτροπής, εν γέννη είχαν την άποψη ότι είναι σημαντικό να ενημερωθούν, να εξυγχρονθούν οι ορισμοί στην οδηγία για την ασφάλεια των προϊόντων και θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τους ε, ορισμούς του νέου νομοθετικού πλαισίου, επειδή η οδηγία για την ασφάλεια των προϊόντων είναι παλαιότερη και κατά κάποιο τρόπο το νέο νομοθετικό πλαίσιο είναι πιο φρέσκο, πιο ενημερωμένο, ειδικά όσον αφορά τους οικονομικούς ε, operators, ε, οι οποίοι ενέχονται άμεσα στις υποχρεώσεις. Και αυτό μας οδήγησε στη διαπίστωση ότι ορισμένε χώρε μέλη χρησιμοποιούν αποκλειστικά τους ορισμούς του νέου νομοθετικού πλαισίου σήμερα και όχι της οδηγίας. Επίσης εξετάσαμε τους ορισμούς του λεγόμενου σοβαρού κινδύνου και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι αντί να τεθεί το ερώτημα για το πώς ορίζεται κατ' ουσία ο σοβαρός κίνδυνος, είναι περισσότερο ένα θέμα αξιολόγησης του κινδύνου και πώς ε, διενεργείται, γίνεται η αξιολόγηση του κίνδυνου. Ε, στο πλαίσιο της Οδηγίας για την Ασφάλεια των Προϊόντων υπάρχουν κατευθυντήριε ε, γραμμέ της RAPEX και υπάρχουν εδώ διάφορε γνώμε για τη χρησιμότητά τη. Ορισμένοι θεωρούν ότι θα είναι βήμα προ τα μπρο, ενώ άλλοι θεωρούν ότι είναι υπερβολικά πλατιά ή άλλοι θεωρούν ότι είναι υπερβολικά ειδικοί. Υπάρχουν λοιπόν διάφορε εκτιμήσει εδώ. Επίση, συμφωνήσαμε στο ότι δεν υπάρχουν ξεκάθαρε κατευθυντήριε γραμμέ όσον αφορά την αξιολόγηση κινδύνου για ενεργοποιημένα προϊόντα. Και αυτό οδήγησε σε κάποιε ανησυχίε ε, εκ μέρου των διαφερόμενων όσον αφορά την δυνατότητα των κατευθυντήριων γραμμών ε, της Εράπεξ για να οδηγήσουν σε, μια, σε ένα συνεπή ορισμό και αξιολόγηση των κινδύνων ε, στο επίπεδο των χωρών μελών. Έγιναν κάποιε προτάσει ευθυγράμμιση ω συμπέρασμα τη μελέτη μα και πρόκειται για δύο βασικά τρόπου όπου η οδηγία για την ασφάλεια των προϊόντων και το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα μπορούσαν να ευθυγραμμιστούν. Μία δυνατότητα είναι να συμπεριληφθούν οι διατάξει για την ε, εποπτεία τη αγορά, τη οδηγία για την ασφάλεια των προϊόντων στο νέο νομοθετικό πλαίσιο και η άλλη δυνατότητα είναι να ενημερωθεί η οδηγία για την ασφάλεια προϊόντων υπό την έννοια να συμπεριλάβει τι σημαντικέ διατάξει, σημαντικότερε διατάξει του νέου νομοθετικού πλαισίου. Και υπάρχουν κάποιε συγκεκριμένε προτάσει ευθυγράμμισης που αφορούν ε, καταρχήν ορισμούς, όπω σας προανέφερα. Θα πρέπει να υπάρξει ευθυγράμμιση ε, των ορισμών, της οδηγίας και του νέου νομοθετικού πλαισίου, ιδιαίτερα όσον αφορά τους οικονομικούς operators ε, και της διάθεσης στην αγορά, τον ορισμό της διάθεσης στην αγορά. Τώρα, άλλες προτάσεις ευθυγράμμισης περιλαμβάνουν τη διευκρίνηση της μεθόδου αξιολόγησης κινδύνου για τον μη καταναλωτικό τομέα και υπάρχουν εδώ κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για τα εναρμονισμένα προϊόντα που δεν είναι καταναλωτικά προϊόντα. Επίσης, όσον αφορά τις υποχρεώσεις των οικονομικών operators, ένα θέμα το οποίο ανέκυψε σε διάφορες συνεντεύξεις είναι το ζήτημα της ανιχνευσιμότητας. Και πολλοί ενδιαφερομένοι είπαν ότι η ανιχνευσιμότητα εξηγείται καλύτερα στο νέο νομοθετικό πλαίσιο. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι σε πολλές χώρες μέλη η ανιχνευσιμότητα, οι ορισμοί της ανιχνευσιμότητας, οι διατάξεις για την ανιχνευσιμότητα ε, συμπεριλαμβάνονται στην ε, εθνική νομοθεσία που μεταγράφει την οδηγία και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν εξετάζουμε την ανάγκη ευθυγράμμισης. Τώρα, όσον αφορά τα δικαιώματα και υποχρώσεις των εθνικών αρχών, το νέο νομοθετικό πλαίσιο και ο κανονισμός 765 περιλαμβάνει το αίτημα για τις χώρες μέλη να εκπονήσουν προγράμματα εποπτείας της αγοράς. Αυτή δεν είναι μια υποχρέωση ρητή στην οδηγία για την ασφάλεια των προϊόντων, όπου λέει ότι μερικά προγράμματα ενδεχομένως θα μπορούσαν να εκπονηθούν. Αυτή είναι μια από τις προτάσεις μας για ευθυγράμμιση. Τώρα, για τα τρία άλλα θέματα τα οποία εξετάσαμε καταρχήν όσον αφορά κοινέ ε, δράσεις για την εποπτεία της αγοράς. Το βασικό ερώτημα αφορούσε τους περιορισμούς που έχουν οι χώρε μέλη να συμμετάσχουν σε τέτοιε δράσει για την εποπτεία τη αγορά, αλλά επίση εξετάσαμε του παράγοντε επιτυχίε και είδαμε τι καθιστά αυτέ τι δραστηριότητε ε, εποπτεία τη αγορά, κοινέ δραστηριότητε, πετυχημένε. Φαίνεται ότι το να υπάρχει, υπάρχουν κοινού στόχου του συμμετέχοντε εξασφαλίζει την επιτυχία. Επίση, η συνεργασία μεταξύ των αρχών εποπτεία τη αγορά ένα παράδειγμα κοινέ δραστηριότητε για τις ε, ομπρέλες ε, ε, στα σολάρια. Επίσης η κατάρτιση του προσωπικού της υπηρεσίας για την εποπτεία της αγοράς και επίσης κοινέ δράσεις δουν τη δυνατότητα περικοπών ή οικονομιών μάλλον, συγγνώμη, ε, σε σχέση με τον τεχνικό εξοπλισμό και σε σχέση με κοινή δοκιμή προϊόντων σε ένα μόνο εργαστήριο. Οι βασικοί περιορισμοί για τις χώρες μέλη να συμμετάσχουν στις κοινέ δράσεις ήταν ε, καταρχήν ε, οι περιορισμένοι πόροι. Πολύ συχνά οι χώρες μέλη πρέπει να δώσουν την προτεραιότητα σε εθνικέ δραστηριότητε, να διαλέξουν μεταξύ των δύο. Πολύ συχνά προτιμούν τι εθνικέ δραστηριότητε από τι κοινέ δράσει Κατά δεύτερο λόγο υπάρχει μεγάλο διοικητικό άχθος που συνδέεται με την υποβολή αιτήσεων για χρηματοδότηση και αναφορά στη συνέχεια που έχει κανείς έχει λάβει τα κονδύλια, όλα αυτά είναι χρονοβόρα και θεωρούνται παχθή. Τέλος υπάρχουν θέματα όπως ε, κάποια χρονοδιαγράμματα που δεν ταιριάζουν με το εθνικό προγραμματισμό ή το θέμα μιας κοινή δράσης δεν θεωρείται σημαντικό για όλες τις χώρες μέλη και υπάρχουν και κάποια γλωσσικά προβλήματα όταν οι αρχές εποπτείας της αγοράς δεν έχουν τις απαιτούμενες γλωσσικές δεξιότητες για να συμμετάσχουν στις κοινέ δράσεις. Επίσης, είδαμε κατά πόσο υπάρχει μια ανάγκη για την εποπτεία της αγοράς που συνδέεται με καταναλωτικά προϊόντα. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σε αυτά τα καταναλωτικά προϊόντα που συνδέονται με το χρήστη. βασική διαφορά είναι εδώ, συνδέεται με το χρήστη και η ικανότητα του χρήστη να κατανοήσει του κινδύνου που συνδέονται με τα διάφορα προϊόντα. Αυτό το οποίο διαπιστώσαμε είναι ότι ένα σημαντικό τμήμα τη εποπτεία αγορά, σύμφωνα με τι χώρε μέλη, απευθύνεται σε καταναλωτικά προϊόντα. Ορισμένοι ενεχόμενοι θεωρούν ότι δεν είναι αναγκαίο να υπάρξει ειδική νομοθεσία εδώ. Αλλά υπήρχαν άλλοι ενεχόμενοι οι οποίοι είπαν ότι είναι αναγκαία η εποπτεία της αγοράς, θεώρησαν ότι είναι απαραίτητη δεν υπήρξε λοιπόν συμφωνία μεταξύ των ενεχόμενων των ενδιαφερόμενων κατά πόσο είναι αναγκαία ή όχι. Τέλος, ένα από τα θέματά μας ήταν η εποπτεία της αγοράς των προϊόντων online και κατά πόσο η φυστάμενη νομοθεσία ε, καλύπτει την ασφάλεια των προϊόντων ε, που αγοράζονται online. Η φυστάμενη νομοθεσία είδαμε ότι πράγματι καλύπτει την ασφάλεια των προϊόντων που αγοράζονται online και οι ενδιαφερόμενοι δεν θεωρούν ότι υπάρχει ανάγκη αναθεώρηση τη φεστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα online προϊόντα. Επίση, υπάρχει οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο που θέτει επιπλέον περιορισμού για τι online πωλήσει και απευθύνεται βεβαίω στις υπηρεσίε, αλλά σε κάποιο βαθμό αφορά και τα προϊόντα. Τώρα, μία πρόταση η οποία προέρχεται από τους είναι ότι πρότεινα ο ρόλος, ε, σχέση με το ρόλο και τον, ε, του των τελωνικών αρχών θα πρέπει να διευρυνθεί. Αυτά είναι τα συμπεράσματά μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κούν. 12 λεπτά διάρκεια παρουσίαση σας. Τέλεια. Είχαμε προγραμματίσει έτσι να ακούσουμε τους δύο επόμενους ε, που θα κάνουν τις παρουσιάσεις πριν να ακούσουμε σχόλια από τους ε, βουλευτές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξέρει καλά η Επιτροπή τον επόμενο. Οι επόμενοι δύο είναι γνωστοί. Και οι δύο εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πού? Πού κάθεται ο επόμενος. Καλώς θα δώσω το λόγο στον κύριο Στέφανο Σόρο που είναι επικεφαλής μονάδας μονάδα τη Γενικής Διευθύνσης ΣΑΝΚΟ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και την Επιτροπή σας που ενδιαφέρεται και πάλι για ζητήματα που σχετίζονται με την εποπτεία της αγοράς ε, για τα καταναλωτικά προϊόντα. Σύντομα, θα ήθελα να θέσω το πλαίσιο. Είχα μία παρουσίαση κάπου που πρέπει να είναι εμφανή στην οθόνη. Πρώτα απ' όλα θα δείτε πως υπάρχει αντίγραφο της έκθεσης ε, της ε, Κομισιόν ε, που παρουσιάσαμε πριν από δύο χρόνια για την εφαρμογή της Οδηγίας για την Ασφάλεια των Προϊόντων, η οποία περιγράφεται ως ισχυρό εργαλείο για το υψηλό επίπεδο προστασία των καταναλωτών, βοήθησε να ανοιχνεύσουμε και να αποσύρουμε χιλιάδες μη ασφαλή προϊόντα από την ευρωπαϊκή αγορά. Νομίζω πως ε, μπορώ να πω πως ποτέ πριν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές δεν είχαν τόσα πολλά και ασφαλή προϊόντα και πουθενά αλλού στον κόσμο δεν υπάρχει ένα σύστημα ενσωμάτωσης ε, διαφόρων χωρών ε, σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο προστασίας ε, των καταναλωτών και ενιαία εποπτεία της αγοράς. Παρ' όλα αυτά, όπως είχε πει και η κυρία Κούνεβα, δεν υπάρχει βεβαίως ποτέ τέλος αυτή η διαδικασία, πάντα μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Βεβαίως ε, ταιριάζει στον σκοπό του στο σύστημα. Υπάρχουν τρόποι να βελτιωθεί. Το δεύτερο στοιχείο που μας παρακίνησε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία αυτή εξέτασης αντικτύπου πιθανής αναθεώρησης της οδηγίας είναι η εμπειρία με 7 ετών εφαρμογής της μαζί με τους συναδέλφους στα κράτη-μέλη μέσω των καθημερινών επαφών μαζί τους στην ε, Επιτροπή για την Οδηγία με τους ενδιαφερομένους έχουμε δει πως υπάρχουν κάποιοι τομείς που θα αναφέρω σε κάνα δύο λεπτά και όπου μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα πιο απλά, πιο ξεκάθαρα και πιο αποτελεσματικά. Ο τρίτος παράγων που μας έβαλε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία είναι πως έχει αλλάξει το ρυθμιστικό πλαίσιο από πρώτης πρώτου φέτος. Η κυρία Κούνεβα είχε αναφέρει το διαφορετικό πλέον το οποίο Έχουμε το νέο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο αποτελείται από την απόφαση 768 του 2008. Ο συνάδελφός μου, ο κύριος Μακμίλαν, ευθυγραμμίζει τις οδηγίες αυτές εναρμόνισης προϊόντων με τις διατάξεις αυτής της απόφασης. Εσείς οι νομοθέτες μας είπατε πως εάν έχουμε νέα νομοθεσία εναρμόνισης ε, των προϊόντων θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις κατήρες γραμμές εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος. Εμείς θεωρούμε λοιπόν πως όσον αφορά τις επιχειρήσεις και την ιχνηλασιμότητα οι διατάξεις απόφασης 768 αξίζουν να ρίξουμε μία ματιά στο πλαίσιο πιθανής αναθεώρησης της οδηγίας. Υπάρχει η απόφαση, ο κανονισμός 765-2008 στο άρθρο 40 λέει πως η Κομισιόν το 2014 το αργότερα θα πρέπει να συντάξει μία έκθεση ή μία πρόταση ενοποίησης για να δούμε πώς βαίνει η ενοποίηση των διάφορων μέσων όλα αυτά τα λέει το άρθρο 40 πέρα λοιπόν από το νέο νομοθετικό πλαίσιο από την θέση ενισχύ της οδηγίας για την ασφάλεια των προϊόντων, αλλά μέσα είναι η ενισχυμένη συνεργασία, ο κανονισμός 2006-2004. Έχουμε έτσι αναπτύξει νέα εργαλεία ενισχυμένης συνεργασία με τα, συνεργασίας με τα κράτη-μέλη. Με όλα αυτά λοιπόν ως δεδομένο αποφασίσαμε να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε το σύστημα καλύτερο, σαφέστερο και όπως σας δείχνει η επόμενη διαφάνεια βασικός στόχος του εγχειρήματος είναι να έχουμε απλούστερους, ξεκάθαρους κανόνες για πιο αποτελεσματική επιτήρηση και εποπτεία της αγοράς. Νομίζω αυτό είναι το κλειδί εδώ πέρα. Δεν επικεντρωνόμαστε σε αυστηρότερους κανόνες για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, όπως η κυρία Κλούζε, όσον αφορά τα μη εναρμονισμένα προϊόντα, η Γενική Οδηγία για την Ασφάλεια των Προϊόντων είναι ένα δίκτυο ασφαλείας και έτσι θα πρέπει να παραμείνει. Η κυρία Σαλτεμόζε ανέφερε, αναφέρατε τα προϊόντα που απευθύνονται σε παιδιά. Επίσης θα μπορούσαμε να έχουμε μια γενική διάταξη για τους χημικούς κινδύνους. Όλα αυτά αφορούν συγκεκριμένα μέσα, η γενική οδηγία για την ασφάλεια των προϊόντων ορίζει την ε, κατηγορία χρηστών και εδώ πέρα ορίζει ειδικά τα παιδιά και τους ηλικιωμένους. Νομίζω μπορούμε να αναφέρουμε επίσης τους ανθρώπους με αναπηρίες. Δεν ξέρω εάν πρέπει να αποτελέσει τώρα ειδικό μέσο για διάφορες κατηγορίες. Το σκεφτικό είναι να έχουμε καλύτερο συντονισμό της δράσης των αρχών των κρατών μελών, ίσους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις και μια εσωτερική αγορά με ασφαλή αγαθά για τους καταναλωτές. Για να σας πω τώρα ποια ήταν η απάντηση των επιχειρήσεων όσον αφορά την επιτήρηση της αγοράς, εμείς συμφωνούμε πως στο ότι οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρηση πρέπει βεβαίω να σημαίνει ενιαία αντιμετώπιση της αγοράς, επίσης όσον αφορά τα επαγγελματικά προϊόντα είναι κάτι που θα το πει ο Ζων Μακμίλαν, αλλά γιατί να έχει άλλους κανόνες η κουδουνίστρα από την πιπίλα. Εγώ δεν βλέπω καμία διαφορά μεταξύ της Γενικής την Ασφάλεια των Προϊόντων και του νέου νομοθετικού πλαισίου. Οπότε θα πρέπει να είναι ενιαία η κατάσταση. Δεν βιαζόμαστε. Θα θα κάνουμε τα πράγματα με την ησυχία μας, συμβουλευόμαστε τους ενδιαφερομένους για τα εξής ζητήματα ειδικά. Πρώτα απ' όλα, τυποποιημένη εντολή με τη Γενική Οδηγία για την Ασφάλεια των Προϊόντων, η οποία είναι η βασική οδηγία εναρμόνιση για οτιδήποτε δεν εναρμονίζει η κοινωτική νομοθεσία Έχουμε προδιαγραφές για προϊόντα από τα τσιγάρα, τους αναπτήρες, οδηγό, ναι, εξοπλισμό όπως τα λεξίπτωτα, ποδήλατα κτλ. Το θέμα είναι πως η διαδικασία είναι μάκρος και ελέστατη και μπερδεμένη και δεν υπάρχει εγγύηση πώς αντιμετωπίζει τις τεχνολογικές εξελίξεις και την πραγματικότητα στην αγορά. Το δεύτερο θέμα το οποίο θεωρούμε πως πρέπει να έχει βελτιώσει είναι τα λεγόμενα μέτρα εκτάκτου ανάγκης του άρθρου 13 καθώς δεν υπάρχει βεβαιότητα για τις επιχειρήσεις. Τα μέτρα αυτά είναι προσωρινά και προσωρινά θα πρέπει να είναι. Μπορούν να οριστούν καλύτερα και να συνδεθούν με μόνιμες λύσεις ε, στην νομοθεσία. Διαφορέ τώρα στην αξιολόγηση ασφαλείας μεμονωμένων προϊόντων και συντονισμό των κρατών μελών. Δεν θα σα κάνω κήρυγμα. Όσοι ήσασταν ε, τις προάλλες στο πρόγευμα της ε, Business Europe Ακούσατε τα αφεντικό μιας ε, μεσαίας Ολλανδικής επιχείρησης ε, που παράγει παιχνίδια που μας έδειξε ένα προϊόν που είχε συναντήσει που είχε τελείως διαφορετικά αποτελέσματα σε διαφορετικές χώρες. Υπήρχε άλλο πρόβλημα στην Ολλανδία, ένα άλλο πρόβλημα στην Ισπανία και ένα πρόβλημα με τα μικρά εξαρτήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε θα θέλαμε να είμαι πιο αποτελεσματική στο να συνεργάζονται οι αρχές των κρατών μελών, να καθίσουν μεταφορικά και να δουν ποιο είναι το πρόβλημα για να προστατεύονται οι καταναλωτές. και να υπάρχει ίση προστασία όσον αφορά το δικαίωμα του καταναλωτή για μια πραγματική εσωτερική αγορά. Και μετά αναφέρω το ζήτημα των ελαφρώς διαφορετικών καθεστώτων επιτήρησης για εναρμονισμένα και μη προϊόντα. Τώρα την επόμενη διαφάνεια μπορούμε να την προσπεράσουμε, γιατί τα κάλυψα ήδη. Τελευταία διαφάνεια αφορά την, τις διαδικασίες. Έχουμε ξεκινήσει μια αξιολόγηση αντικτύπου, όπως είναι και σωστό. Συμβουλευόμαστε όλους τους ενδιαφερομένους, έχουμε δημόσια διαβούλευση. Σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη απάντησαν και στηρίζουν τους στόχους μας σχεδόν ομόφωνα. κατοπίν θετικό. Έχουμε καλές και διαφορετικές απαντήσεις από τις επιχειρήσεις, τις ενώσεις, ε, τα επεξεργαζόμαστε και θα επανέλθουμε και εδώ και στα κρατη Τους ακούμε. Λοιπόν, 1η Δεκεμβρίου εδώ στις Βρυξέλλες θα έχουμε μία διάσκεψη των ενδιαφερομένων για την αναθεώρηση της Γενικής Οδηγίας για την Ασφάλεια των Προϊόντων και για το αποτέλεσμα τη δημοσία διαβούλευση. Θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. very Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρήσιμα αυτά τα οποία μας είπατε και από ό,τι κατάλαβα θεωρείτε πως πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση για να απλοποιηθεί η Γενική Διεύθυνση Ασφάλεια των Θα δώσω τον λόγο στον επόμενο μιλητή, ο οποίος επίσης είναι γνωστός στην Επιτροπή μας, ο κύριος Ζακ Μακμίλαν έχει τον λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι, έχω την αίσθηση πως έχω ξανάρθει εδώ και έχω, τα έχω ξαναζήσει αυτά. Και ευχαριστώ την γραμματεία που δεν βρήκε μια αυτογραφία μου. Λοιπόν, το νέο νομοθετικό πλαίσιο υιοθετήθηκε τον Ιούλιο, 9 Ιουλίου. Είχαμε έναν κανονισμό στην οποία αναφέρθηκε ο Στέφανος. Έχουμε δύο συμπληρωματικούς στόχους. Ο κανονισμός θα ορίσει το γενικό πλαίσιο και τους άμεσα εφαρμοστέρους κανόνες για την πιστοποίηση και την επιτήρηση της αγοράς, ενώ η απόφαση προσπαθεί να εναρμονίσει και την νομοθεσία και τις εθνικές πρακτικές σε πράγματα όπως δημοσιεύσεις κατασκευαστών, διανομέων κτλ. Η εφαρμογή λοιπόν της εποπτείας αγοράς σημαίνει πρώτα απ' όλα να παρακολουθούμε τα κράτη-μέλη στα μέτρα που λαμβάνουν για να εφαρμόσουν τον οργανισμό, αλλά επίσης σημαίνει μέσω μακροπρόθεσμη παρακολούθηση των κρατών μελών, γιατί η επιτήρηση της αγοράς δεν είναι κάτι που ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου φέτος και σταμάτησε την 2η Ιανουαρίου, είναι μια συνεχής διαδικασία. Οπότε ο βαθμός εποπτείας αγοράς θα αλλάξει όπως αλλάζει και η κατάσταση. Οπότε είναι και αυτό ένα μέσο μακροπρόθεσμο έργο. Σημαίνει πως η εφαρμογή του κεφαλαίου 3 του κανονισμού περιέχει το εξή σημαντικό. Το κεφάλαιο εποπτείας της αγοράς συμπεριλαμβάνει τα ελεγχόμενα προϊόντα από τρίτες χώρες, δηλαδή ο έλεγχος προϊόντων από τρίτες χώρες είναι κομμάτι της εποπτείας αγοράς. Και μετά, όπως ο Στέφανος ήδη είπε, σύμφωνα με την απόφαση 768, ευθυγραμμίζουμε την νέα νομοθεσία με την απόφαση, ενσωματώνουμε τους ορισμούς, τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων κατασκευαστών για να υπάρχει μια συνοχή η αδυναμία της απόφασης έγκυται στο ότι νομικά μιλώντας δεν μπορούμε να την επιβάλλουμε μέχρι να συμπεριληφθούν οι διατάξεις σε νομοθεσία. Αλλά τι συμβαίνει. Χρησιμοποιούν πολύ την οδηγία ως έχει και πολλά κράτη-μέλη εργάζονται με βάση αυτές τις διατάξεις. Η εφαρμογή άμεσα σημαίνει πως τα κράτη-μέλη έπρεπε να κάνουν πολλή δουλειά. Έπρεπε να βρουν τις αρμόδιες εθνικές αρχές, εθνικές, τοπικές κτλ. Να τα πούν όλα αυτά στην Κομισιόν και στα άλλα κράτη-μέλη. Αυτό το έχουν κάνει όλα τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν αυτά στο site της Κομισιόν. Έπρεπε επίσης να συντάξουν εθνικά προγράμματα υποπτήρες αγοράς για το 2010 Όλα τα κράτη-μέλη έχουν προγράμματα για το 2010. Ένα είναι ένα πολύ γενικό. 12 είναι τομεακά και 14 είναι μεικτά. Επίσης όλα περιέχουν κυρώσεις και διατάξεις προβλέψεις για το σηματάκι CE και τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν πει πως έχουν ήδη διατάξει στην εθνική νομοθεσία για τις κυρώσεις. Οπότε, όπως βλέπετε, συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα, έχουμε δηλαδή πάρα πολλές πληροφορίες που βεβαίως θα πρέπει να εξετάσουμε γιατί δεν είναι πράγματα τα οποία ξέραμε χρειαστεί χρόνος να επεξεργαστούμε αυτές τις πληροφορίες. Τα κράτη-μέλη επίσης είπαν ξεκάθαρα πως είδαν τις διατάξεις και το τι ισχύει στην εθνική του νομοθεσία. 18 κράτη-μέλη είπαν πως θα επιφέρουν σοβαρές αλλαγές στην νομοθεσία, 12 έχουν ορίσει διυπουργικούς συντονιστές Βεβαίω αυτό σημαίνει πως και οι υπόλοιποι είχαν και τα υπόλοιπα 15, οπότε τώρα όλα τα κρατημέλη έχουν διυπουργικούς συντονιστές. Κατά το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον είναι και δείχνει τη σημασία του κανονισμού για την εποπτεία προϊόντων τρίτων χωρών, 17 κρατη έχουν ορίσει ειδικού συντονιστέ μεταξύ των αρχών υποτεία αγορά και των τελωνίων κάτι το εξαιρετικά θετικό. Και νέα κράτη-μέλη ανακοινώνουν βαθύτατες αναδιαρθρώσεις του μηχανισμού εποπτείας αγοράς. Εφαρμογή από την Κομισιόν τώρα. Ο κανονισμός αναφέρεται στη χρήση του RAPEX. Είμαστε σε μια διαδικασία στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΡΑΠΕΞ. Προσπαθούμε να ενσωματώσουμε τα στοιχεία που απαιτεί ο Το άρθρο 23 μας λέει πως θα πρέπει να έχουμε μια βάση δεδομένων για την υποπτήρια της αγοράς γενικώ. Εμείς πάντα είπαμε πως θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε την υπάρχουσα βάση δεδομένων, την ICSMS, που δημιουργήθηκε από τα κράτη-μέλη. Διαπραγματευόμαστε τη συγκεκριμένη σύμβαση. Υπάρχει η βάση δεδομένων, το θέμα είναι πώς θα μπει στο νομικό πλαίσιο της Ένωσης. Εν τω μεταξύ βεβαίως υπάρχουν ενδιάμεση κανόνες επικοινωνίας που λειτουργούν αρκετά καλά. Απλά είναι λίγο πιο πολύπλοκο το θέμα από το να είχαμε την ε, λύση της πληροφορικής. Ξεκινήσαμε με κάποιον συντονισμό όπως απαιτεί ο κανονισμός Αυτό το οποίο κάναμε κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών είναι να συντονίσουμε το πώς συντάσσουν τα προγράμματα τα εθνικά εποπτείας αγοράς. Φτιάξαμε λοιπόν ένα υπόδειγμα. Δυστυχώς το υπόδειγμα αυτό εγκρίθηκε κάπως αργά το 2009 οπότε πολλά κρατημέλη δεν μπόρεσαν να το ακολουθήσουν αλλά αναμένουμε να το ακολουθήσουν τα κρατη στο μέλλον. Οπότε θα μπορέσουμε να συγκρίνουμε τι κάνουν το κρατη σε ποιους τομείς και να δούμε αν μπορέσουμε να έχουμε προτεραιότητες της Ένωσης και όχι εθνικές. Και εκεί πέρα θα δούμε πού χρειαζόμαστε συντονισμό, κοινέ δράσει και παρέμβαση της κοινότητας. τελευταίο σημείο εδώ πέρα αναφέρεται συντονισμό των αρχών εποπτείας αγοράς και των τελωνίων. Αλλά καθώς είναι εδώ πέρα η κυρία Εμπειρία από την Γενική Διεύθυνση Τελωνίων, θα εξηγήσει εκείνον νομίζω το συντονισμό αυτών. Πού βρίσκομαι. Α, ναι. Η φύση των υποχρεώσεων σύμφωνα με τον κανονισμό είναι πολύ σοβαρέ υποχρεώσει. Πρώτα απ' όλα υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να οργανώσουν την αγορά. Έτσι λέει ο κανονισμό. Τα κράτη μέλη θα οργανώσουν την εποπτεία τη αγορά. Δεύτερον, τα υποχρεώνουν να δράσουν. Όχι μόνο να οργανώσουν την εποπτεία τη αγορά, αλλά πρέπει προληπτικά να ασκούν έλεγχο και να αντιδρούν όταν βλέπουν μη ασφαλή προϊόντα. Και πρέπει να έχουν τα μέσα να επιβάλλουν διορθωτικές δράσεις ή ακόμα και να καταστρέψουν προϊόντα. Ο κανονισμός ισχύει πέρα από την υγιεινή και την ασφάλεια των καταναλωτών αφορά όλη την νομοθεσία που καλύπτει υγιεινή, ασφάλεια περιβάλλον, ε, ασφάλεια πόρου εργασίας, Επίσης, η υποχρέωση στα κράτη-μέλη συμπεριλαμβάνει ένα πονηρό άρθρο που υποχρεώνει τα κράτη-μέλη όχι μόνο να έχουν την αρμοδιότητα, αλλά και τα μέσα να τα κάνουν αυτά. Η υποχρέωση να έχουν την αρμοδιότητα σημαίνει πως οι επιθεωρητές πρέπει να έχουν την αρμοδιότητα να λάβουν απόφαση σε σχέση με το προϊόν και να μην περιμένουν τα δικαστήρια κτλ για να αποσύρουν το προϊόν από την αγορά. Έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν τα κρατη μέλη και την Κομισιόν και να συντονιστούν εσωτερικά με όλες τις εθνικές αρχές και τα τελωνία και με τα άλλα κράτη-μέλη. Ένα τελευταίο σημείο πολύ σημαντικό ο κανονισμός στηρίζει τομεακή νομοθεσία και υπάρχει μια, διαδικασία παρακολούθησης των επικίνδυνων προϊόντων. Δηλαδή, εάν δούμε ένα προϊόν το οποίο είναι επικίνδυνο σε ένα κράτος μέλος, όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη πρέπει να λάβουν παρόμοια δράση. Οι σχέσεις τώρα με την Γενική Οδηγία για την Ασφαλεία των Προϊόντων δεν θα πω πάρα πολλά, τα ανεφέρει ο συνάδελφος. Αυτό το οποίο θα έλεγα είναι πως πρώτον δουλεύουμε με βάση λέξη σπεσιάλη και κατά περίπτωση κρίνουμε που ισχύει το κείμενο. Υπάρχει το κείμενο των διαφορετικών πεδίων εφαρμογής γιατί είναι ευρύτερος ο κανονισμός, δηλαδή πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσουν οι ειδοποιήσεις RAPEX και η παρακολούθηση, η συνέχεια που θα δοθεί, καθώς είναι διαφορετικά τα πράγματα, η διατάξει στην οδηγία από ό,τι στον κανονισμό. Τι σημαίνουν αυτές οι διαφορές. Μπορούμε να το δούμε αυτό και να πούμε πως εντάξει δεν είναι τόσο διαφορετική ορισμοί, αλλά το κείμενο διαφέρει. Το ένα είναι η οδηγία και το άλλο είναι κανονισμός. Και σύμφωνα με τη Γενική Οδηγία για την Ασφάλεια των Προϊόντων, οι επιχείρησει και οι οργανώσει καταναλωτών δεν έχουν αρμοδιότητες. Έχουμε όμως εμείς αρμοδιότητες σύμφωνα με τον ε, κανονισμό, οπότε μπορούν να πάνε στι εθνικέ αρχές στα δικαστήρια. Οπότε οι διαφορέ είναι πιο σημαντικές από όσο φαίνονται. Γιατί αν ακολουθήσουμε τη μία οδό ε, είμαστε στο πλαίσιο της οδηγίας, ενώ με την άλλη είμαστε στα εθνικά δικαστήρια κατά των εθνικών αρχών. Οπότε είναι σημαντικές οι συνέπειες. Και το θέμα είναι θα πρέπει να έχουμε δύο συστήματα ή όχι. Δεν το ξέρω. Πολλά μέλη έδειξαν πως θέλουν να τα εφαρμόσουν όλα αυτά. Είναι σαφές πως θέλουν ένα σύστημα, πολλά προσπαθούν να το εφαρμόσουν ως ένα σύστημα, αλλά γνωρίζοντας πως αυτό θα έχει συνέπειες. Οπότε θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά, αλλά η αίσθησή μου είναι πως πρέπει να ενημερώσουμε την οδηγία, να ευθυγραμμιστεί, αλλιώς θα καταλήξουμε δύο διαφορετικά συστήματα. Δεν ναι, θα πάω στο τελευταίο. Τα χρόνια, εδώ, εδώ και χρόνια πάμε από εδώ και από εκεί. Είχαμε την πρώτη οδηγία, μετά είχαμε την αποσυράπεξ, ε, προχωρούσαμε με γρήγορα άλματα. Και τώρα έχουμε το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Κάνουμε πάντα άλματα. Η συνύπαρξη τώρα των δύο κειμένων θέτει το ερώτημα του τι θα κάνουμε σε σχέση με την εποπτεία της αγοράς και το μήνυμα είναι πως το μήνυμα που λαμβάνουμε είναι πως τα κράτη-μέλη και οι επιχειρήσεις είναι ένα απλό σύστημα γιατί ε, είναι σαφέστερο έτσι και ξέρουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και είναι ευκολότερο να το εφαρμόσουν και οι εθνικές αρχές γιατί το να είναι απλό το σύστημα έχει χρήσιμο και για τις εθνικές αρχές. Ευχαριστούμε κύριε Μακμέλαν. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι ήταν ιδιαίτερο χρήσιμο για μένα αλλά και για μας εδώ να ακούσουμε ότι η εφαρμογή του πακέτου για τα αγαθά βελτιώνεται και αυτό είναι πολύ θετικό. Πριν από ένα χρόνο μας, είπαν, μας είπε η Rumble ότι έχει αντιμετωπίσει προβλήματα, ενώ τώρα μας, είπατε, μας λέτε ότι η κατάσταση βελτιώνεται. Χαίρομαι πάρα πολύ που τόσο εσύ, εσείς όσο και ο κύριος Σόρο θεωρείτε ότι χρειάζεται μια αναθεώρηση, δηλαδή υπάρχει μια ενιαία άποψη μεταξύ των δύο γενικών διευθύνσεων. Ίσως θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για το πώς θα πρέπει να γίνει, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που και οι δύο συμφωνείτε ότι χρειάζεται ένα είδος αναθεώρησης. Ήταν πολύ χρήσιμο λοιπόν. Τώρα θα ήθελα να καλέσω τα μέλη εδώ να θέσουν ερωτήματα ή να κάνουν σχόλια. Παρακαλώ. Η πρώτη είναι η κυρία Χάνσλικ. Ναι. Ε, επιτρέψατε μου να θέσω δύο ερωτήσεις. Τη μία εκ μέρους της συγγήτρης κυρίας Κοχόλη που δυστυχώς δεν τα κατάφερε να έρθει σήμερα εδώ. Η κυρία Κοργόλα ήθελε να ξέρει ποια είναι η βασική διαφορά στην ε, δοκιμή και παρακολούθηση καταναλωτικών και μη καταναλωτικών προϊόντων. Εσείς ε, πιστεύετε ότι αυτές οι δύο κατηγορίες προϊόντων θα μπορούσαν να συνδυαστούν και να αντιμετωπιστούν κοινά, ως κοινέ. Και αν ισχύει κάτι τέτοιο, ποιο θα ήταν το πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης και ποιες θα ήταν οι προκλήσεις που συνδέονται με μια τέτοιου είδους προσέγγιση. Δηλαδή το να συνδυάσει κανείς τη Γενική Οδηγία για την Ασφάλεια Προϊόντων και το κανονισμό για την επι... της αγοράς. Ένα άλλο ερώτημα εκ μέρους της Επιτροπής ΣΥΝΤΕΡ. Μία ερώτηση προς την Επιτροπή. Η Γενική Διεύθυνση ΣΕΝΚΟ ε, εκπώνησε το σύστημα RAPEX το οποίο χρησιμοποιείται από αυτή την Γενική Διεύθυνση για να παράσχει στις κινέζικες ε, αρχές κάποια στοιχεία όσον αφορά τα προϊόντα αυτά που προέρχονται από την Κίνα και τα οποία θεωρούνται, αναγνωρίζονται στην Ευρώπη ως επικίνδυνα και κατά συνέπεια αποσύρθηκαν από την ευρωπαϊκή αγορά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν πώς λειτουργεί ακριβώς αυτό το σύστημα λειτουργεί εύρυθμα κατά την άποψή σας ή θεωρείτε ότι κάποια αντίστοιχα συστήματα θα πρέπει να, να δημιουργηθούν, να συσταθούν και για άλλους εμπορικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα εκείνους τους εταίρους που κατασκευάζουν ε, προϊόντα τα οποία δεν εμπίπτουν στο σύστημα RAPEX. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η επόμενη κυρία Σάιλερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τους ομιλητές. Η ερώτησή μου αφορά το θέμα της χρηματοδότησης. Και θα ήθελα να πω, σε σχέση με το τελευταίο ομιλή, όταν αναφέρεται στα μέσα που πρέπει να, αξιοποιηθούν. Νομίζω ότι εννοείται οικονομικά μέσα. Ε, τώρα υπάρχουν τέτοιες ε, περικοπές στον προϋπολογισμό της Μεγάλης Βρετανίας, τόσο μεγάλες περικοπές ε, στο δημόσιο τομέα, που νομίζω ότι θα έχει μια επίπτωση στις δυνατότητες εποπτείας της αγοράς. Στη σελίδα 9 της έκθεσης του Κοινοβουλίου λέει ότι υπάρχουν κάποια εμπόδια, κάποιοι φραγμοί στη συμμετοχή των χωρών μελών που συνδέονται με τη χρηματοδότηση. Θα ήθελα να μα σχολιάσετε σχετικά. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλή ερώτηση. Καταρχήν, ε, πιστεύω ότι η πρώτη ερώτηση επικεντρώνεται, ε, απευθύνεται μάλλον στον κύριο Σόρο και η δεύτερη στον κύριο Μακμίλαν. Αλλά και οι δύο μπορείτε να απαντήσετε. Κύριε Σόρο, θέλετε να απαντήσετε στην κυρία Χάνσλε. Ναι. Ε, πραγματικά είναι, η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Ε, η Rapex ε, China λειτουργεί πολύ καλά, ε, δεν στοιχίζει τίποτα και έχουμε πολλά στοιχεία. Έχουμε εκατοντάδες εξαγωγικές άδειε που ανακαλούνται από τις κινέζικες αρχές στη βάση πληροφοριών που τους δώσαμε μέσω του συστήματος RAPEX της Κίνας. Έχουμε ε, πάρα πολλές ε, δράσεις που ανέλαβαν οι κινέζικες αρχές, γιατί το κινέζικο σύστημα έχει ως εξής. Αν θέλετε να έχετε μια νόμιμη εξαγωγή, χρειάζεται μια άδεια εξαγωγής από την κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν μας δίνει ένα ενίο σημείο επαφής με τις κινέζικες αρχές. Το δεύτερο, η δεύτερη πιο σημαντική επίπτωση της RAPEX Κίνα είναι ότι έχει μια άμεση επίπτωση γιατί ήταν κίνητρο για τις κινέζικες αρχές να ξεπεράσουν τα όρια της, του απλού συστήματος κοινοποίησης, γνωστοποίησης, ε, προχωρώντας σε μια πιο αυστηρή εποπτεία της αγοράς, ιδιαίτερα όσον αφορά τον τομέα των παιχνιδιών. Και αναφέρουμε στο 2007, όπου χιλιάδες ε, εγκαταστάσεις επιθεωρήθηκαν, ορισμένες έκλεισαν και ορισμένες εξαγωγές άδειες ανακλήθηκαν. Τώρα, θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε λεπτομερή έκθεση ε, παρακολούθηση από τις αρχές κάθε τρεις μήνες. Έχουμε διάφορες ε, αναφορές ερευνών που γίνονται με διάφορες τροποποίησεις. Ε, είναι μια σχέση πραγματικά που θα πρέπει να συνεχίσει. Ε, η πολιτική εμπλοκή είναι ε, θετική. Θα συναντήσουμε τον Κινέζο Υπουργό σε μερικού ε, μήνε και ο κύριο Χάρμπουρ θα συμμετάσχει σε αυτή την αποστολή, σε την επίσκεψη. Νομίζω ότι όπως καταστήσαμε αρκετά σαφές προηγουμένως, το πλαίσιο για την ε, επιτήρηση της αγοράς μπορεί να επωφεληθεί από την ε, ομοιομορφία, από την ομογενοποίηση. Η υγεία και η ασφάλεια των καταναλωτών είναι ένας πολύ σημαντικός ε, στόχος της πολιτικής μας. Νομίζω ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε την ε, προσπάθειά μας όσον αφορά το θέμα αυτό της ε, ασφάλειας. Τώρα για την κυρία Στάιλ, κατά πόσο οι περικοπές στον προπολογισμό θα έχουν μια επίπτωση. Προσωπικά αυτή είναι η άποψή μου και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό επιτροπές όπως η ΙΜΚΟ να χτυπάνε στις πόρτες των κρατών μελών και τα πιέζουν για εφαρμογή των ε, νόμων. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν κανόνες για συνεργασία οι οποίοι κανόνες θα επιτρέπουν και σε εμά και στα κράτη-μέλη ε, να μπορούμε να έχουμε την αναγκαία υποστήριξη. Θα πρέπει λοιπόν να μην λησμονούμε ότι έχουμε καλούς κανόνες, καλύτεροι κανόνες είναι καλοί, αλλά καλύτερη εφαρμογή των υφισταμένων κανόνων είναι ακόμα πιο σημαντικό θέμα και ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να λιπάνουμε το σύστημα, για να φτιάξουμε πραγματικό δίκτυο αρχών, είναι κάτι ευπρόσδεκτο και ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο στις παρούσες συγκυρίες. Σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ σαφής η απάντηση. Κύριος Μακμίλαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω δύο σχόλια να κάνω. Το πρώτο αφορά το θέμα των δοκιμών. Η δοκιμή ενός προϊόντος καταναλωτού ή προϊόντος μη καταναλωτού είναι παρόμοιο. Το θέμα είναι η ένταση, ε, πόσο τακτικά γίνονται οι δοκιμές, ποια στοιχεία θα πρέπει να δοκιμάζονται σε σχέση με τους ενδεχόμενους χρήστε ενό ε, προϊόντος. Η ίδια η δοκιμή δεν επηρεάζεται, αλλά οι προϋποθέσεις που τίθεται για τη δοκιμή αυτές κάνουν τη διαφορά και γι' αυτό έχουμε συγκεκριμένους κανόνες ε, που αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα. Και σε κάποιες περιπτώσεις οι απαιτήσει για προϊόντα καταναλωτού είναι αυστηρότερε από ότι για άλλα προϊόντα. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν αλλάζει η δοκιμή. Τώρα, το άλλο θέμα της χρηματοδοτήσεως, το σκοτσέζικο αίμα μου ε, παγώνει πάνω σε αυτό το θέμα, αναπηδά και ανατριχιάζει. Δεν έχουμε άρθρο στον κανονισμό που να λέει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διαθέτουν τα μέσα θα πρέπει να το καταλάβετε, είναι πρωτοπού αυτό. Πρέπει να καταλάβετε ότι δεν είναι η αρχή υποπτία της αγοράς που έχει το πρόβλημα, δημιουργεί το πρόβλημα για την εξέβρεση μέσων. Αυτές οι αρχές, οι εποπτικές, ουρλιάζουν, θέλουν πόρους και δεν τους δίνουν. Δεν έρχονται οι πόροι από τον κεντρικό προϋπολογισμό. Ο κανονισμός αυτός θα έχει αποτελέσματα αν όλοι έχουν τον τρόπο και τα μέσα να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται τα χρήματα και να έχουν, διαθέτουν οι υποπτικές αρχές περισσότερα μέσα. Συμφωνώ με τον Στέφανο. Υπάρχουν όρια. Πρώτα απ' όλα έχουμε τις περικοπές του προϋπολογισμού. Πρέπει να πολεμήσουμε τις περικοπές του προϋπολογισμού και απ' την άλλη άλλες πολιτικές προτεραιότητες. Όλοι έχουμε διαφορετικές προτεραιότητες. Και θα πρέπει να εξισορροπηθούν. Η εποπτεία της αγοράς δεν είναι από τα πιο σεξι θέματα που βρίσκονται στην πολιτική αρένα το, τις μέρες μας. Όχι, δυστυχώς. Δεν κερδίζει κανείς τις εκλογές με καλή εποπτεία της αγοράς. Κυρία Ρούλε, ε, συγγνώμη δεν σας είδα πριν, έχετε το λόγο. Κανένα πρόβλημα. Δεν πειράζει. Θα ξεκινούσαμε με τις περικοπές του προϋπολογισμού που ξεκίνησαν πριν από την κρίση όταν συζητούσαμε τότε το πακέτο, διαπιστώσαμε πως δεν υπάρχει αρκετός προϋπολογισμός για την επιτήρηση της αγοράς. Το ερώτημά μου είναι τώρα, αυτά τα πρότυπα που είπατε, τι επίδραση θα έχουν. Το πρόβλημά μας είναι πως στο ευρωπαϊκό επίπεδο ως βουλευτές δεν έχουμε κάποιο μέτρο σύγκρισης μεταξύ της υποπτίας αγοράς στα διάφορα κράτη-μέλη. Δεν ξέρουμε τι γίνεται, γιατί δεν έχουμε πολλά δεδομένα. Και νομίζω πως αυτό το υπόδειγμα θα ε, καθιστούσε πιο διάφανη την κατάσταση. Επίσης κάποια κράτη-μέλη έχουν αποκεντρωμένη διοίκηση και είναι ακόμη πιο δύσκολο να ξέρουμε αν υπάρχει ασφαλής επιτήρηση και αποτελεσματική. Το ένα είναι αυτό. Πώς θα έχουμε αυτή τη διαφάνεια είναι κάτι το οποίο έχει υπερκύψει. Μπορώ να πω πως στη δική μου τη χώρα έχουμε συνεχώς προβλήματα με την οδηγία της συσκευασίας, με τα παιχνίδια και συχνά δεν επιτυχαίνει η υποπτία της αγοράς. Αλλά λένε πως η ευρωπαϊκή νομοθεσία παρά το... και δεν καταλαβαίνει ο κόσμος πως η ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει κάνει τα περισσότερα στον τομέα αυτών. Δεύτερον, Ράμπολ, δεν καταλαβαίνω πώς καταλήξατε το συμπέρασμα πως οι διαφορετικοί ορισμοί δεν αποτελούν πρόβλημα για την επιτήρηση της αγοράς. Με κλείσει λίγο αυτό. Δεν ξέρω πού βασιστήκατε. Εγώ ξέρω από τη Γερμανία πως λόγω αυτών των διαφορών υπάρχουν διαφορετικές οδηγίες χρήσης. Και όταν υπάρχουν βεβαίω διαφορετικέ οδηγίε χρήση, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα πρακτική εφαρμογή τη εποπτεία αγορά. Οπότε θα ήθελα να μάθω πώ καταλήξατε εσεί σε αυτό το συμπέρασμα. Ευχαριστώ κυρία Ρούλε. Πρώτα απ' όλα, κυρία αν θέλετε να σχολιάσετε αυτά που είπε η κυρία Ρούλε. Και μετά συνεχίζουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά το θέμα τα προγράμματα τα εθνικά για την εποπτεία της αγοράς όταν συνεργαζόμαστε με τις εθνικές αρχές να καταλήξουμε σε κάποιο πρότυπο Είχαμε επίγνωση του προβλήματο των πληροφοριών. Είναι σαφέ ότι από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουμε να μπορούμε να δίνουμε τι περισσότερε δυνατέ πληροφορίε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διότι νομίζουμε ότι όσον αφορά αυτό είμαστε σύμμαχοι. Και καμιά φορά ίσω να έχετε περισσότερη επιρροή από ότι εμεί. Άρα όλοι κερδίζουν επωφελές για όλους. Έχουμε άλλο πρόβλημα. Δεν μπορούμε αυτές τις πληροφορίε να τις δημοσιεύουμε ευρέως. Αν αρχίζει κανείς να δημοσιεύει το ποια εθνική αρχή πρόκειται να κάνει ποιου ελέγχου επί ποιων προϊόντων και πότε, τότε τι να πω. Αν δώσουμε αυτές τις ε, πληροφορίες αυτοπυροβολούμεθα, διότι και άλλοι θα παίρνουν τις πληροφορίες. Ξέρω ότι δεν εννοούσατε αυτό αλλά έχουμε ένα πρόβλημα μέχρι ποιο βαθμού μπορούμε να προχωρήσουμε όσον αφορά τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών και συμφωνήσαμε με τι εθνικέ αρχέ ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δημοσιεύουμε όσο δυνατόν περισσότερε πληροφορίε, αλλά εντό ορίων, να μην προειδοποιούμε του ελεγχόμενου. Είναι σαν την ταινία Κάτσι 22, ένα φαύλο κύκλο δηλαδή. Η αποκέντρωση. Τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικές καταστάσεις Κάποιοι έχουν κεντρικό σύστημα, αλλά λιγότερο κεντρικό. Εμείς στην Βρετανία έχουμε 220 αρχές, οι Γερμανοί έχουν τα γερμανικά ομόσπονδα κρατήδια κλπ. Εδώ τίθεται το θέμα της υποχρέωσης συντονισμού, εσωτερικού συντονισμού. Εκεί πρέπει να γίνει διαφορά. Και εκεί θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρον να δούμε πόσα κράτη-μέλη έχουν εφαρμόσει τους μηχανισμούς συντονισμού, διότι είναι ο μόνος τρόπος που μπορούν να χειριστούν την κατάσταση μόνα τους. Ο κανονισμός κατά κάποιο τρόπο βοηθάει τι εθνικέ αρχές να αναδομηθούν και να ελέγχουν περισσότερο τι δραστηριότητε του. Αλλά αυτό δεν θα γίνει εν μία ανοιχτή. Χρειαστεί χρόνο. Κυρία Κούν, ευχαριστώ. Κυρία Ρούλε, όπως είπα, οι εμπλεκόμενοι θεωρούν ότι θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν οι ορισμοί, υπάρχουν διαφορές, αλλά είπαμε ότι μπορούμε να τις ξεπεράσουμε. Μπορούμε να, συνεργα... να τις περάσουμε, τις δυσκολίες, για να μην βλάψουμε την εποπτεία της αγοράς και την ασφάλεια των προϊόντων. Ένα κάτι άλλο που ανέκυψε είναι ότι η, οδηγία, η Γενική Οδηγία για την ε, ε, τον έχω των προϊόντων ερμηνεύεται με διαφορετικό, για την ασφάλεια των προϊόντων ε, ερμηνεύεται με ποικιλόμορφο τρόπο στα διάφορα κριτημέλη και πιστεύω ότι αυτό απαντάει. Ο κ. Κρόιτσμαν είναι ο τελευταίος από το γύρο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις. Καταρχήν αναφέρθηκε η δικτύωση των διαφόρων IT συστημάτων. Πότε θα προχωρήσουμε εδώ, γιατί νομίζω ότι αυτό θα συνιστούσε μεγάλη πρόοδο ε, σε σχέση με την ε, αποκέντρωση, το σχεδιασμό της ε, αγοράς, της παρακολούθησης της αγοράς με τον κεντρικό έλεγχο. Το δεύτερο ερώτημα είναι το πώς θα τα καταφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν λέει ότι οι χώρες μέλη είναι υπεύθυνε οι αρμόδιες για την οργάνωση της επιτήρησης της αγοράς πώς ε, θα αλλάξει αυτή η κατάσταση. Ε, έχετε μία ιδέα ε, σε σχέση με την δομή της επιτήρησης της αγοράς. Πώς θα επενδύσει κανείς αυτή τη δομή, που υπάρχουν οι αδυναμίες και αν υπάρχουν κάποιες αδυναμίες ή ελλείψεις, πώς θα προσπαθήσει, πώς θα τα καταφέρει η Κομισιόν να τις ξεπεράσει. Ευχαριστώ κύριε Κρόιτσμαν. Βλέπω και το επόμενο θέμα για την αποκτή τη αγορά. Αυτό βλέπω να διαφέρει τι ερωτήσει. Το θέμα είναι να πάμε κατευθείαν σε αυτού που θα μιλήσουν το θέμα. Α λάβετε υπόψη τι ερωτήσει του κ. Κρόιτσμαν και μετά ξαναδούμε το λόγο στον κύριο Σόρο και τον Ζακ Μακμίλεν. Ε, εν συντομία. Σχόλιο έχω. Όσον αφορά αυτά που είπε η κυρία Κούντ. Οι εμπορευόμενοι λένε ότι οι διαφορετικοί ορισμοί και το παιδεία δεν είναι τόσο σημαντικά, μπορούν να τα καταφέρουν. Διότι με προσανατολισμού και λοιπά, κατευθείας γραμμέ μπορούν να τα καταφέρουν. Πράγματι ισχύει αυτό. Αλλά δεν κατάλαβαν όλοι τι συνέπειε της διαφοράς μεταξύ οδηγία και κανονισμού. Τα περισσότερα κράτη μέσα σε αυτό το τομέα έχουν συνηθίσει τι οδηγίε. Άρα συνήθισαν πολιτικέ συμφωνίε διαπραγματεύσει για την εφαρμογή. Με κανονισμό όμω, η κανόνα του παιχνιδιού είναι εντελώ διαφορετική. Τα δικαστήρια και δεν υπάρχει διαπραγμάτευση. Αυτό δεν το έχουν πιάσει ακόμα. Ε, ότι οι διαφορές μπορούν να κάνουν τη διαφορά λόγω των διαφορετικών νομικών συνεπιών. Πολλοί εμπλεκόμενοι φορείς δεν το έχουν καταλάβει ακόμα και πολλέ εθνικέ αρχές δεν το κατάλαβαν αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα πάμε στο επόμενο τμήμα. Ρίτσαρντ Λόσον, επικεφαλής του κλάδου τεχνικών κανονισμών για τις ε, τεχνικές δεξιότητες ε, του Ηνωμένου Βασιλείου. Καλημέρα όλοι, σε όλους σας. Ευχαριστώ κυρία μου. Ευχαριστώ πολύ για την δυνατότητα που δίνετε στον Ηνωμένο Βασίλειο συμμετάσχει στο εργαστήριό σας. Πρώτη διαφάνεια παρακαλώ. Δεν θα χρονοτριβήσω, επί του θέματος, δείχνει όμως την κατανομή των ευθυνών στο Ηνωμένο Βασίλειο, κόκκινο στο κέντρο αφορά την νομοθεσία, το λευκό στο κέντρο είναι οι βαθικές, βασικές αρμόδιες αρχές που διαπραγματεύονται και εφαρμόζουν ε, την ε, οργανωτική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και το, το μπλε δείχνει τις αρχές εποπτήσεις της αγοράς και τα άσπρα κουτάκια δείχνουν τα κομμάτια της νομοθεσίας για τα οποία είναι υπεύθυνα τα διάφορα ε, υπεύθυνε οι διάφορε αρχέ που είναι στο μπλε. Μπορείτε να διαβάσετε με την ησυχία σα μετά το διαγραμμά. Θέλω να προχωρήσω. Κοιτάξτε τι ερωτήσει που έχετε θέσει. Ε, κοίταξα τι ερωτήσει. Πιέζει ο χρόνο, θα είμαι σύντομο και θα αναφέρω μόνο κάποια συγκεκριμένα και στι ερωταπαντήσει μπαίνουμε σε λεπτομέρειε. Προκλήσει για τι αρχέ εποπτεία τη αγορά Καταρχά, το να αποφασίσει κανεί ποιο, μοντέλο θα, ποιο μοντέλο θα ακολουθήσει για την εποπτεία τη αγορά και στα πλαίσια τη επικουρικότητα θα πρέπει να ασχοληθεί με θέματα αν πρωταρχικά θα εστιάζεται επί τη παιδεία ή επί τη εφαρμογή, ε, πόσο είναι σχεδιασμένο έλεγχο αγορά, πόσο είναι έλεγχο ανταποκρίσει διαμαρτυρίε θα βασίζεται στην αξιολόγηση του κινδύνου ή ευρεία κλίμακα δειγματοληψία, ποιε είναι οι προτεραιότητε, η επι τη εφαρμογη ποσο ειναι σχεδιασμενο ελεγχο αγορα ποσο ειναι ελεγχο ενταποκρισει διαμαρτυριε θα βασιζεται στην αξιολογηση του κινδυνου η ευρεια κλιμακα δειγματοληψια ποιε ειναι οι προτεραιοτητε η ασφαλεια ισότιμε συνθήκες στην εσωτερική αγορά. Κάποια άλλη πρόκληση είναι η δυνατότητα να μοιράζεται κανείς πληροφορίε για εξολόγηση των κινδύνων και να πληρώνει και να, να οδηγείται στη σωστή κατανομή των πόρων. Μετά συνεργασία μεταξύ των διαφόρων φορέων, διαφορετικές προτεραιότητε των διαφόρων φορέων, διαφορετική τρόπη συνεργασία και να μην ε, οι προμηθευτές να μην πιέζονται. Βεβαίως η περιπλοκότητα των προϊόντων, η τεχνολογική που αυξάνεται, το αυξανόμενο κόστος των δοκιμών και η έλλειψη τεχνογνωσίας είναι μόνο κάποιοι φορείς που μπορούν να σας πούνε κατά πόσο υπάρχει συμμόρφωση ενός προϊόντος με τους κανόνες ή όχι και να έχουν συμμετάσχει στην ανάπτυξη του προϊόντος και βεβαίως από ό,τι μας είπαν και όλο και περισσότερα προϊόντα έρχονται από τέτοιε χώρε. Γενικά η ροή των προϊόντων και όσο και περισσότερη οικονομική ε, φορείς εμπλέκονται στην, ε, στα προϊόντα, εμπλέκεται η αλυσίδα και είναι και ποιοι έχουν τι ευθύνε. Αυτοί που κατασκευάζουν τα προϊόντα, αυτοί που τα εισαγάγουν, αυτοί τα διανέμουν. Και θα πρέπει να μην υπάρχει και καλυμμένο ε, προστατευτισμό. Θα πρέπει να είναι ελεύθερη αγορά και να μην δημιουργούμε φραγμού στο εμπόριο τεχνική φύσεω ή άλλη φύσεω. Μετά την επόμενη διαφάνεια, καλέ πρακτικέ, με τι πρακτικέ, θα πρέπει να γνωρίσουμε ότι οι περισσότερε επιχειρήσει θέλουν να συμμορφώνονται με τον νόμο. Και ο καλύτερο τρόπο να το κάνουν αυτό είναι να εκπαιδευτούν και να ξέρουν επιχειρήσει νομικέ υποχρεώσει. Θα πρέπει να ανταποκρινόμεθα στι νόμιμε διαμαρτυρίε για μη συμμόρφωση από διάφορε επιχειρήσει που διαμαρτύρονται και καιρό, αλλά μην παρεμβαίνουμε στην ίδια την αγορά. Δεν θα πρέπει να γίνουμε το μέσο για προστατευτισμό. Θα πρέπει το αντιθυμιστικό βάρο να είναι το ελάχιστο δυνατό, συμβατό βέβαια με το υψηλό επίπεδο συμμόρφωση. Θα πρέπει οι επιχειρήσεις να καταβάλουν προσπάθειες ούτω ώστε να υπάρχει εσωτερική, ε, εσωτερικός ελέγχος για την παραγωγή και συνεργασία με άλλους φορείς εντός κρατών μελών όλο και πιο σημαντικό μεταξύ κρατών μελών να υπάρχει συνεργασία και να ανταλλάσσονται οι εμπειρίες. Τώρα στην επόμενη διαφάνεια πάμε. Με ενδιαφέρεται το θέμα της συνεργασίας μεταξύ των αρχών τελωνίων, των τελωνιακών αρχών και των αρχών εποπτείας της αγοράς. Εμείς παραδοσιακά έχουμε καλή εμπειρία στον αφορά αυτό τη συνεργασία των δύο φορέων εισοδήματα και ε, τελωνία. Δηλαδή, τελωνία και υποπτικές αρχές. Ήταν πιο περιορισμένα εκτός Αγγλίας, αλλά ακολουθούμε τις σωστές δεώσεις διαβιβάσεις και η Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχου της Αγοράς έχει δημιουργηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, περιμένοντας ότι την εφαρμογή της 76-52-8 και πρέπει να γίνεται αυξανόμενη η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών και των τελωνίων και μεταξύ των φορέων των ίδιων των εποπτικών αρχών. Θα πρέπει να γίνεται ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών μεταξύ των φορέων όσον αφορά και στα πλαίσια τη επιτροπή Συντονισμού τη αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα βάλουμε νομική προστασία όσον αφορά τη ροή από τα τελωνία πληροφοριών από τα τελωνία προ τι εποπτικέ αρχέ, για να, διατη... να προστατεύσουμε τα εμπορικά μυστικά. Και στον Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζουμε τη σημασία που έχουν τα τελωνία 20, τη συνεργασία σε επίπεδο ευρωπαϊκή Ενώση μεταξύ τελωνίων και υποπτικών αρχών. Θα σα ενδιαφέρει και το θέμα τη ανιχνευσιμότητας και της online, των online αγορών. Ανιχνευσιμότητα είναι θέμα όλο πιο σημαντικό, γιατί είναι σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον η ροή των προϊόντων και ασχολούμεθα με αυτό, προσπαθούμε να το λύσουμε μέσω συνεργασίας με τους ε, εισαγωγείς, τους χονδρεμπόρους και τους λιανεμπόρους. Θέλουμε να συνεργαστούμε, διότι η αγοραστική δύναμη είναι ένα σκυλό ε, εργαλείο για συμμόρφωση. Εάν οι λιανοπολιτές θέλουν να κρατήσουν τη φήμη τους για να πολλούν και προϊόντα που συμμορφώνονται με τους ε, νόμους. Η αγορά online είναι πρόκληση. Και οι αρχέ στο Ηνωμένο Βασίλειο μαθαίνουν διάφορε αρχέ η μία από την άλλη και προοδεύουν τεχνικέ του. Στην Επιτροπή Συντονισμού γίνεται ανταλλαγή και βασικοί φορεί όπως το eBay θέλουν να βοηθήσουν. Τα προϊόντα που παρέχονται θέλουν να συμμορφώνονται με τον νόμο. Όσον αφορά την εχνησιμότητα, πιστεύουμε ότι το πακέτο ευθυγράμμισης, δηλαδή η απόφαση 768-28 να εφαρμόζεται, είναι κάτι που ε, θα συντονίζει τα καθήκοντα που υπέχουν η παραγωγή, εισαγωγή και διανομή. Νομίζω ότι τήρησα το χρονοδιάγραμμα. Θα σταματήσω εδώ και μετά θα προβώ σε άλλα σχόλια στην ανταλλαγή των απόψεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα επόμενος ομιλητής, Γιάν Κόνικ, πρόεδρος της ProSafe και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Και ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε στο εργαστήριο αυτό. Πιθανότατα μπορούμε να περάσουμε την πρώτη διαφάνεια, η οποία δεν είναι και τόσο ενδιαφέρουσα. Το μόνο πράγμα που πρέπει να θυμόσαστε από την πρώτη διαφάνεια είναι ότι είμαι υπεύθυνο ε, κράτου μέλου για την εποπτεία τη αγορά. Δουλεύω για τι βελικέ αρχέ, αλλά είμαι εδώ σαν πρόεδρο του ProSafe. Για εσά που δεν ξέρετε τι είναι το ProSafe, να σα δώσω μια σύντομη παρουσίαση σε ένα λεπτό, να σα εξηγήσω τι κάνει αυτό ο φορέα, γιατί είμαι εδώ. Και πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Η ProSafe είναι, βλέπετε, είναι για, για την εφαρμογή των κανόνων για τα ασφαλή προϊόντα. Δημιουργήθηκε το 1990 και χρησιμοποιείται σε μια βάση, σε μια πλατφόρμα για ανταλλαγή πληροφοριών και σε μια βάση για ευρωπαϊκά προγράμματα και για το συντονισμό κοινών δράσεων. Στόχος ε, του φορέα μας είναι να προωθεί ανεπίσημες συζητήσεις και διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών και των υπαλλήλων των αρχών αυτών ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών και βελτίωση εν γέννη της εποπτής αγοράς όσον αφορά τα προϊόντα, την ασφάλεια των προϊόντων στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο. Χρειάζεται να λέμε ποιο είναι ο στόχο μα. Ποιο είναι ο στόχο μα, να διευκολύνουμε τη συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών για να βελτιώνονται τα προϊόντα, η ασφάλεια των προϊόντων και η ασφάλεια των υπηρεσιών. Άρα, βλέπετε, είναι περίεργη η κατάσταση που αντιμετωπίζω εγώ. Είμαι υπεύθυνο για την εποπτεία τη αγορά ενό κράτου μέλου, αλλά δεν μιλώ για το κράτο μέλο μου, ούτε για την αρχή την οποία εκπροσωπώ, ε, στην οποία δουλεύω. Εκπροσωπώ Ευρωπαϊκό Οργανισμό, που είναι ένα οργανισμό ο οποίο δεν απαρτίζεται από τα κράτη-μέλη συγκεκριμένα, αλλά από εκείνου που εργάζονται στον τομέα. Ό,τι πω εδώ δεν είναι δεσμευτικό για το κράτο μέλο μου, ούτε κανένα άλλο κράτο μέλο. Αλλά έχω μεγάλη εμπειρία όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς στην Ευρώπη. Λοιπόν, η εποπτεία της αγοράς. Ετέθησαν κάποια ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις για τις αρχές, τις εποπτικές. Πρώτα απ' όλα, να σας πω το εξή. Ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις. Θα πρέπει να θυμόμαστε πρώτα ποιος είναι ο στόχος της εποπτείας της αγοράς. Ποιος είναι ο στόχος. Επόμενη διαφάνεια. Βεβαίως. Έχουμε πολλαπλούς στόχους πρέπει να ξέρουμε ότι στην αγορά διατίθεται μόνο ασφαλή προϊόντα. Αυτό είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών. Επίσης, θέλουμε να ισχύουν ισότιμες συνθήκες στην αγορά. Κάθε κατασκευαστής, παραγωγός, διανομέας πρέπει να πληρεί τις ίδιες προϋποθέσεις, έχει τις υποχρεώσεις αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον τομέα, για τη βιομηχανία. Και εξασφαλίζουμε και τους δύο προαναφερθέντες στόχους, συνεπάγεται ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων επίσης. Δείτε λοιπόν ποιε είναι οι βασικές προκλήσεις για την εποπτεία της αγοράς και τις ε, εποπτικές αρχές. Υπάρχει μια πρόκληση όσον αφορά τη συνεπή ερμηνεία κάποιων πραγμάτων. Πρώτα απ' όλα των ορισμών. Τα προβλήματα δεν είναι ξεπέραστα. Οι διαφορέ μεταξύ των ορισμών καμιά φορά είναι μικρή, πολύ μικρή, αλλά μπορεί να δημιουργεί προβλήματα στην πράξη. Πιο συγκεκριμένα η διάθεση στην αγορά είναι κάτι που μπορούμε να συζητούμε επί ώρε. Είναι... Όταν μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπαίνει στην αγορά. Όταν πάει στο κατάστημα, όταν στην αποθήκη, όταν είναι στα ράφια. Τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικέ απόψεις. Τουλάχιστον οι υποπτικέ αρχέ έχουν διαφορετικέ απόψει. Άλλο θέμα είναι η ερμηνεία των υποχρεώσεων. Υποχρεώσεις για τους κατασκευαστές, τους διανομής, παραγωγούς. Τρίτον, ερμηνεία του κινδύνου. Ποιος είναι ο σοβαρός κίνδυνος. Έχουμε αρκετά εργαλεία για να προσπαθήσουμε να εναρμονίσουμε, αν μπορώ να το πω αυτό, αυτό το τομέα, αλλά απομένουν ακόμα κάποιοι πολιτισμικοί φραγμοί πολιτισμικές τάσει και προκαταλήψουν όσον αφορά την αξιολόγηση του κινδύνου. διαφορέ αντιλήψεων. Προαναφέρθηκε ότι η βασική πρόκληση για τι αρχές μας είναι οι πόροι. Όχι μόνο οικονομικοί πόροι, αλλά και τεχνικοί πόροι. Και μάλλον στελέχη, πώς προσωπικό. Ποικίλει από κράτο μέσο σε κράτο μέλο. Αν λείπουν οι ανθρώπινοι πόροι, αλλού λείπουν περισσότερο ανθρώπινοι πόροι, αλλού περισσότερο τα χρήματα, συνήθω λείπουν και τα δύο. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι οι δυνατότητες δοκιμών είναι και αυτό μια πρόκληση για μας. Δεν έχουν όλα τα κράτη-μέλη τις ίδιες δυνατότητες για δοκιμές. Οπότε έτσι φτάνουμε στην επόμενη διαφάνεια που λέει ποιες είναι οι καλές πρακτικές. Πρώτα απ' όλα καλή πρακτική κατά την άποψή μου είναι να συνεργάζονται τα κράτη-μέλη, να μοιράζονται και να ομαδοποιούν τους πόρους. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω κοινών δράσεων, όπου τα κράτη-μέλη μπορούν να ομαδοποιούν τις τεχνικές δυνατότητες, ανθρώπινους πόρους, τα χρήματα. Είδαμε στα αποτελέσματα προγράμματος. Το Διπούκ, ένα, έχουμε ένα, το EMAS δημιούργησε ένα βιβλίο για την εποπτεία της αγοράς Ένα αποτελέσμα του προγράμματος ήταν ένα φόρουμ για γρήγορες συμβουλές. Υπάρχει δυνατότητα οι αρχές, οι υπάλληλοι των εποπτικών αρχών να συνομιλήσουν με συναδέλφους τους ανεπίσημα ε, για να ζητήσουν κάποιες πληροφορίες για ένα προϊόν. Ένα προϊόν που αξιολογείται έχουμε αποθηκευμένες γνώσεις και μπορούν ανεπίσημα να είναι προσβάσιμες αυτές οι γνώσεις με αυτόν τον τρόπο. Ε, καλή πρακτική είναι τα διάφορα προγράμματα, ε, ε, εθνικά προγράμματα εποπτής αγοράς να δημοσιοποιούνται χωρίς να αναφέρεται συγκεκριμένα πού, πώς και πότε θα γίνονται οι ελέγχοι. Αλλά πρώτα πρέπει να ενημερώνονται τα εμπλεκόμενα μέρη, μετά να προειδοποιούνται και μετά προσπαθείς να επιβάλλεις το νόμο. Είναι πολύ πιο αποτελεσματικό να ενημερώνεις κάποιον και αν δεν το κάνει αυτό που πρέπει, τότε να βγεις και να πας να προσπαθήσεις να τον υποχρεώσεις να το κάνει. Πιο αποτελεσματικό. Η συνεργασία με εξτεριωνιακών αρχών και υποπτικών αρχών είναι προαπαιτούμενο. Ε, το θέμα είναι ότι οι αρχές αυτές δεν έχουν ήδη προτεραιότητες Καμιά φορά υπάρχει έλλειψη γνώσεως, τεχνική γνώση από πλευρά τελωνίων. Εγώ δεν ξέρω από την άλλη πολλά για τα τελωνία, άρα και οι τελωνιακές αρχές δεν ξέρουν και πολλά για την ε, αποτεχνική σκοπιά την ασφάλεια των καταναλωτών. Προσπαθούμε να τους δώσουμε καταλόγους, να δώσουμε πληροφορίες με απλό τρόπο στα τελωνία. Ε, ανάλυση κινδύνου. Δεν, δεν θέλουμε να δούμε ένα επικίνδυνο έχει ένα προϊόν, αλλά αν ένα προϊόν, συγκεκριμένο προϊόν, είδο προϊόντος που προέρχεται από συγκεκριμένη πηγή, μπορεί, θα μπορούσε να είναι ανασφαλές. Αυτό εξαρτάται από την προέλευση, από το είδος του προϊόντος. Θα μπορούσε το τελωνίο να εστιαστεί επί των προϊόντων που εισέρχονται, διότι και οι τελωνιακοί τότε ε, έχουν κάποιους περιορισμένους όρους, Επόρους μάλλον, συγγνώμη. Αυτό που λέω είναι ότι η αποτελεσματική σημαίνει ότι πας κοντά στην πηγή, μπορεί να σταματήσει το προϊόν πριν μπει στην Ευρώπη, τότε είναι η αποτελεσματική προσέγγιση, αλλά για να έχει αποτελέσματα πρέπει να ελέγχει όλα τα κομμάτια τη αλυσίδα, ξεκινώντα με το σχεδιασμό και φτάνοντα μέχρι το προϊόν που πάει στο ράφι. Και όταν γίνεται έλεγχο αγορά στα καταστήματα. Για να κλείσω, ήθελα να πω ότι είναι ανιχνευσιμότητα των προϊόντων online, απαγορεύσει μόνιμε, ε, η ανιχνευσιμότητα προ όφελο όλων, διάθεση στην αγορά είναι σημαντικό τα online προϊόντα δημιουργούν προβλήματα διότι γίνεται ιδιωτική εισαγωγή απ' έξω από την ΕΟΧ. Έρχονται σε πακέτα ε, στον ιδιώτη τα προϊόντα. Μόνιμες απαγορεύσεις, δεν μπορεί να απαγορεύσεις μόνιμα προϊόντα απλά ε, χωρίς ε, να δημιουργήσεις εμπορικούς φραγμούς. Ας πούμε τα καροτσάκια για τα παιδιά ε, ήταν ένα παράδειγμα που μπορούσαμε να βελτιώσουμε τα προϊόντα χωρίς να βάλουμε γενική απαγόρευση. Πρέπει να εναρμονιστούν οι διαδικασίες, να δίνουμε περισσότερους πόρους, αυτά πρέπει να γίνουν, και να υπάρχει εσωτερικός και εξωτερικός συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο κατά μέλλον. Αυτό που χρειάζεται ακόμα, το βλέπουμε στην επόμενη διαφάνεια, είναι η ευρωπαϊκή νομοθεσία για εναρμονισμένες διαδικασίες υπάρχει. Έχουμε τις εθνικές, εθνικούς ελέγχους για επιδόσεις βάση κινδύνου, αλλά χρειάζεται συντονισμός κάπου ανάμεσα όσον αφορά τις διαδικασίες της δράσης και βάση δεδομένων που να μπορεί να χρησιμοποιήσουν οι υποπτικές αρχές. Και για να κλείσω, αν επιτρέπετε, Θέλω να πω ότι αναφέρθηκε ότι δεν μπορεί να κερδίσει κανείς εκλογές με καλή υποπτή της αγοράς, αλλά εγώ πιστεύω ότι σίγουρα μπορεί να χάσει εκλογές με κακή, κακό έλεγχο, κακή υποπτή της αγοράς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Συμφωνώ. πολύ. με αυτό. Ε, συγγνώμη που σας έδωσα τόσο περιορισμένο χρόνο για την ιδιαίτερως ε, χρήσιμη και σημαντική, ιδιαίτερως χρήσιμες και σημαντικές παρουσιάσεις. Θα μπορούσαμε όμως να περάσουμε μέρες να συζητούμε για αυτά τα θέματα. Ωστόσο, στην... το μόνο που θα μπορούσα να πω είναι ότι στην Ολομέλεια τα μέλη έχουν μόνο ένα χρόνο αγόρευση στη διάθεσή τους. Λοιπόν, ο επόμενος ομιλητής ε, είναι από τη Γενική Διεύθυνση Τεξτού αναφέρατε την ανάγκη συνεργασίας. Θα ήθελα να καλωσορίσω την Caroline Εντερή. Thank you very much. I would like to... Ευχαριστώ πολύ. The opportunity to... Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δώσετε την ευκαιρία να πω μερικά λόγια για το ρόλο των τελωνίων για αυτό το σημαντικό τομέα της εποπτείας της αγοράς και της εξασφάλισης της αγοράς. Και θα ήθελα να πω κάποια πράγματα σχέση με τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλυθεί από την Γενική Διεύθυνση. Ήδη επισημάνθηκε ότι οι τελωνιακέ αρχές παίζουν έναν όλο και σημαντικότερο ρόλο στην ε, εποπτεία της αγορά και έχουν ξεκάθαρες ε, υποχρεώσει ε, που εμπίπτουν στον κανονισμό 765. Ε, και ο ρόλος τους ε, εξελίσσεται όλο και περισσότερο προς την ε, προστασία των πολιτών και φεύγει από την επιβολή των φόρων. Λοιπόν, ε, ένας αποτελεσματικός τρόπος εξασφάλισης ελεύθερης κινητικότητας στην αγορά και εξασφάλιση ότι δεν τοποθετούνται μη συμβατά προϊόντα στην αγορά είναι να διενεργούνται έλεγχοι και εδώ τα τελωνία μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο. Αλλά επίσης θα πρέπει να έχουμε κατά νου ένα στόχο της αναθεώρησης των, του περιβάλλοντος των τελωνίων, τον οποίο επεξεργασόμαστε. Δηλαδή να μην παρεμποδίζουμε το νόμιμο εμπόριο, γιατί έχουμε όλο και περισσότερα αιτήματα να εξασφαλίζουμε ούτως ώστε το, οι διεκπαιρεώσεις να γίνονται ταχαίως στα σύνορα, οι εμπορικές διατυπώσεις. Δηλαδή θα πρέπει να βρούμε εδώ μια ισορροπία μεταξύ διευκόλυσης του εμπορίου και εξασφάλισης ε, του καταναλωτού. Θα πρέπει να βρούμε εναρμοσμένους και απλούς ε, ρόλους που αφορούν την εποπτεία της αγοράς. Όσο περισσότερο κινούμεθα προ ένα ενιαίο σύστημα, τόσο καλύτερα είναι τα πράγματα για μα. Η ιδέα μα είναι να αναπτύξουμε μια εναρμονισμένη προσέγγιση για την διενέργεια των τελωνιακών ελέγχων όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων. Γι' αυτό ο κ. Λόσον ανέφερε το ότι η Κομισιόν μαζί με τις τελωνικές αρχές των χωρών μελών δημιούργησαν μια ομάδα προγραμματισμού η οποία εκπονεί κάποιες κατευθυντήρες γραμμές όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων. Και στο πλαίσιο αυτή τη ομάδα, αναγνωρίσαμε τρεις ε, τομείς κλειδί για τις δράσεις μας. Καταρχήν, να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο συνεργασίας μεταξύ τελωνικών αρχών και αγορών. Δεύτερον, να μοιραστούμε βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τη συνεργασία αλλά και την ενέργεια των ελέγχων. Και τέλος, να δημιουργήσουμε μια, έναν εναρμονισμένο έλεγχο και να βελτιώσουμε το management. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένω. Ξεκινήσαμε την εργασία μα το 2008 με ένα πρώτο σεμινάριο όπου συναντήθηκαν οι αρχέ εποπτεία τη αγορά και οι τελωνιακέ αρχέ και εκεί αναγνωρίσαμε την ανάγκη να ληφθούν έντονε ε, δράσει για να αναπτυχθούν αυτοί οι τομεί τη συνεργασία. Ε, Πέρσι συστάθηκε μια ομάδα εργασία, περιλαμβάνει όλε τι χώρε μέλη, συν την Νορβηγία. Οι κύριοι στόχοι του project είναι να βοηθούν τα τελωνία να κατανοήσουν τι νέε του ευθύνε που εμπίπτουν στον κανονισμό, ο οποίο ε, τέθηκε σε ισχύ αυτό το έτο. Επίση, να παρακολουθήσουμε και να αξιολογήσουμε την τρέχουσα κατάσταση σε όλε τι χώρε μέλη. Ορισμένε ε, χώρε είναι πολύ εξελιγμένε όσον αφορά την ανάπτυξη ελέγχων για την εποπτεία τη ε, αγορά και την συνεργασία μεταξύ των διαφόρων αρχών. Και επίσης θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες των τελωνιακών αρχών, οι ανάγκες. Το πρόγραμμα ξεκίνησε πέρσι, έχουμε ήδη, είχαμε ήδη τρεις συναντήσεις, συμφωνήσαμε όσον αφορά τη μέθοδο εργασίας και την διάρθρωση των κατευθυντήριων γραμμών και ελπίζουμε να παρουσιάσουμε την άνοιξη του 2011 τα τελικά αποτελέσματα. Λοιπόν, αναμένουμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των ελέγχων για την ασφάλεια των προϊόντων και επίση ε, να εξασφαλίσουμε ότι οι τελωνικές αρχές μπορούν να αναγνωρίσουν ένα προϊόν ως επικίνδυνο και να μπορούν άμεσα να αναλάβουν κάποια δράση να υπάρχει δηλαδή μια συνεχής ροή ανταλλαγής πληροφοριών. Επίσης θέλουμε να αναπτύξουμε κάποια κριτήρια, κοινά κριτήρια αναγνώρισης κινδύνου στην Τελωνική Ένωση και επίσης να ενημερώνουμε τα δεδομένα και τις πληροφορίες και να επεκτείνουμε τις κατευθυντήρες γραμμές σε διάφορες τομείς προϊόντων που αναγνωρίζονται ως έχοντας ε, ως χρήζουσες, ε, χρήζοντες ε, κάποιας ιδιαίτερης προσοχής όσον αφορά τη διενέργεια ελέγχων. Επίσης, να κοινοποιήσουμε τα αποτελέσματα και να παράσχουμε συνδρομή στις χώρες μέλη όσον αφορά την εφαρμογή ε, των τελωνιακών ελέγχων. Αυτό όσον αφορά την ομάδα του project. Επίσης, θα ήθελα εδώ να προσθέσω δύο σημεία που αφορούν την εργασία στο μέλλον και τα οποία ήδη τέθηκαν εδώ, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να φέρουμε καταρχήν της ε, πωλήσει online, ένα θέμα το οποίο αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία, αλλά και ανησυχίες για τους, τους γιατί η police on sales σημαίνει ε, ότι τα τελωνία θα πρέπει να ασχοληθούν με όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία φτάνουν εκεί, που είναι όλο και περισσότερα, και θα πρέπει να προσαρμόσουν τις μεθόδους εργασίας σε αυτή τη νέα πρόκληση. Και αυτή τη στιγμή ε, αυτή την εποχή οργανώνουμε το Παρίσι την άλλη εβδομάδα ένα σεμινάριο με, τα, με τις ελληνικές αρχές για να δούμε ποιες, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή και ποιες είναι οι βέλτιστες ε, πρακτικές που θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε. Ε, αφορούν θέματα παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά επίσης θέματα διατύπωσης ε, σωστών προδιαγραφών. Ένα άλλο θέμα είναι η αξιοπιστία των τελωνίων. Ε, η, συμβατότητα με τις, συμμόρφωση με τις προδιαγραφές δεν είναι ζήτημα μόνο των δημόσιων αρχών, αλλά και των προμηθευτών. Και θα πρέπει οι προμηθευτές επίσης να συμμορφώνονται. Λοιπόν, θα πρέπει να ε, εξασφαλίσουμε τόσο την διευκόλυνση του εμπορίου αλλά και την ε, αξιοπιστία των ε, προϊόντων. την αξιόπιστη προμήθεια των ε, προϊόντων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ χρήσιμο που ακούσαμε και αυτή την παρουσίαση. Και τώρα θα περάσουμε στους επόμενους δύο μιλητές, που είναι οι τελευταίοι ομιλητές σήμερα. Ο Στίβεν Ράσελ, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας της ΆΝΕΚ και ο οποίος ε, ε, νομίζω θα δώσει και λίγο χρόνο στην Τάνια Βάνεμπεργκ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτή εξ αρχής ότι παρόλο που κάνω την παρουσίαση αυτή εκ μέρους της ΆΝΕΚ, εμείς είμαστε ενωμένοι όσον αφορά την ανάγκη αναθεώρησης της Γενικής Οδηγίας για την Ασφάλεια Προϊόντων. Είμαστε βασική ευρωπαϊκή οργάνωση καταναλωτών. Ε, χαίρομαι υπάρχει ένα συνάδελφο από την ε, Βέλκ, η Σίλβια Νάρ. Ε, νομίζω ότι υπόθηκε ήδη ότι η Γενική Οδηγία για την Ασφάλεια των Προϊόντων υπήρξε μια επιτυχία. Αλλά όπω τα πάντα στη ζωή αυτή επιδέχεται βεβαίω κάποιων βελτιώσεων και αυτή η αναθεώρηση μα δίνει ακριβώ αυτή την ευκαιρία. ευκαιρία Τώρα, όσον αφορά την τυποποίηση, ε, η σχετική έκθεση ε, εγκρίθηκε χθε από την Επιτροπή. Νομίζω ότι τώρα μπορούμε να πάμε στο κρεβάτι μας και να ανερευτούμε για τα δυνατά και τα δύναμα σημεία της ε, τυποποίησης. Έχουμε κάποιες ανησυχίες σε σχέση με την αρχική απόφαση της Κομισιόν που ορίζει τις προδιαγραφές ασφαλείες γιατί αυτή η απόφαση δεν είναι νομικά δεσμευτική. Επίσης, οι οργανώσεις των Ευρωπαίων προδιαγραφών υποδιαγραφών δεν είναι να δεχθούν μια εντολή ευρωπαϊκής τυποποίησης. Και η χρήση είναι θελοντική. Συνεπώς δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι προδιαγραφές αυτές θα εξελιχθούν. Και όσον αφορά το άρθρο 13 και τα έκτακτα μέτρα, αυτό μπορεί να προκαλέσει κάποια σύγχυση ε, μεταξύ των οικονομικών ε, φορέων και των καταναλωτών. Ε, θα πρέπει να υπάρξει μια ανανέωση στο τέλος της περίοδου ισχύω, έστω και αν δεν βρεθεί μια ικανοποιητική λύση όπως είναι νέες ευρωπαϊκές Πιστεύουμε επίσης ότι οι πολιτικές αποφάσεις που έχουν άμεση επίπτωση στην προστασία ευημερία των καταναλωτών θα πρέπει να λαμβάνονται από τους ρυθμιστές σε κοινοτικό επίπεδο ένα παράδειγμα είναι η, τα μηχανήματα ε, μουσικής ε, που έχουν ορισμένα επίπεδα για τον ήχο. Αλλά αυτό δίνει ένα φάσμα, δεν ε, τίθεται ένα απόλυτο επίπεδο στην εντολή. Επιτρέπει σε αυτόν που κάνει την τυποποίηση να θέσει ο ίδιο τα όρια και αυτό θα έπρεπε να επιτρέπεται από τους ρυθμιστές. Επίση, μα προκαλεί ανησυχία η έλλειψη μια διαδικασία ε, ε, ε, ρήτρας διαφύλαξης όπως το άρθρο 13 που δίνει μια δυνατότητα στον καταναλωτή να προσφύγει. Η επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Ε, προτείνουμε το νομοθετικό πλαίσιο για τι ε, απαιτήσει σχεδιασμού για τα ενεργειακά προϊόντα θα πρέπει να λειτουργεί ως μοντέλο για, τα, για την ασφάλεια των προϊόντων. Αυτή η οδηγία ε, εξετάζει ε, την υφέτηση κάποιων μέτρων για συγκεκριμένε κατηγορίε προϊόντων και συμπληρώνεται από ένα φόρουμ διαβούλευση, στο οποίο περιλαμβάνονται όλοι οι ενεχόμενοι, όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Επίσης, προτείνουμε αποτήσεις για προσφυγές όσον αφορά την αναθεώρηση του πλαισίου, οι ευρωπαϊκές ε, προδιαγραφές θα πρέπει να διατυπώνονται μέσω μιας εντολής που δίδεται από την Κομισιόν και υπάρχει βεβαίως μια ανάγκη να ενισχύσει η διαδικασία ευρωπαϊκή τυποποίηση, στην οποία θα συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια δυνατότητα να εφαρμόζονται υψηλότερα, υψηλότεροι τρόποι αξιολόγησης από ό,τι στην παλαιότερη οδηγία. Η οδηγία δεν παρέχει τη δυνατότητα να επιλεγεί το κατάλληλο επίπεδο αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Ε, η οδηγία αφορά όλα τα καταναλωτικά προϊόντα τα οποία δεν καλύπτονται από ειδικέ οδηγίες. Ακόμα και εκείνες ακόμα και εκείνα που θα μπορούσαν να θέτουν ε, σοβαρούς κινδύνους. Σε ορισμένε περιπτώσεις εξασφαλίζεται ένα, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ένα υψηλότερο επίπεδο ε, στη βάση μιας αξιολόγησης κινδύνου. δεν πιστεύουμε ότι με επιστοποίηση μέσω τρίτων λύνεται το πρόβλημα. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να στοχεύει η πιστοποίηση εκεί όπου υπάρχει ένας σημαντικός κίνδυνος. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σφαιρικό πλαίσιο για την ασφάλεια των καταναλωτών τόσο για τα προϊόντα όσο και τις υπηρεσίες. Σήμερα υπάρχει ένα κενό στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όσον αφορά γιατί η ασφάλεια των υπηρεσιών δεν καλύπτεται από καμία ευρωπαϊκή νομοθετική πράξη. Κάθε ορισμένα προϊόντα καλύπτονται από την ειδική και την ασφάλεια. Για παράδειγμα, εξοπλισμός που είναι υπεύθυνο για πολλά ατυχήματα δεν καλύπτεται από την οδηγία. Ε, το ίδιο. Water slides, πώς τα λέμε. Ε, το ίδιο θα μπορούσε να ισχύει και για τις ε, νεροτσουλήθρες, που είναι επικίνδυνα προϊόντα. Ε, θα θέλαμε να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την επιτήρηση της αγοράς. Λέμε ότι είναι δυνατόν να έχουμε του καλύτερου δυνατού νόμου στην Ευρώπη, μπορούμε να έχουμε τι καλύτερε υποδιαγραφέ, αλλά χωρί αποτελεσματική υποπτία τη αγορά και τα δύο αυτά γίνονται άχρηστα. Ναι, υπάρχει η ρύθμιση, ο κανονισμό 765, αλλά ακούσαμε ήδη ε, από μια έκθεση που έγινε ένα χρόνο πριν ε, της Επιτροπής ότι δεν είναι όλες οι χώρες μέλη διατεθειμένες να εφαρμόσουν. Δηλαδή, οι ε, ορισμένες που θέλουν να δεν έχουν τους απαιτούμενους πόρους. Νομίζω ότι η επιτήρηση της αγοράς δεν είναι από τα θέματα που κερδίζουν τις εκλογές και η ισότητα πόρων υπάρχει σε πολλές χώρες. Ο κανονισμός δεν το πρόβλημα των κοινών ορισμών. Η επιτήρηση της αγοράς θα πρέπει να γίνει από κοινού στις διάφορες χώρες μέλη Πιστεύουμε επίση ότι είναι σημαντικό να λαμβάνονται κάποια μέτρα ούτε ώστε να επιτρέπουν μια ταχεία αναγνώριση ελαττωματικών μη ασφαλών προϊόντων. Και στο πλαίσιο αυτό καλούμε την συνεργασία για απαιτήσει όσον αφορά τι υποχρεώσει των κατασκευαστών ε, στο πλαίσιο του νέου νομοθετικού πλαισίου. Και πιστεύουμε ότι τεχνολογίε όπω η ΑΕΦ μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά από την οπτική του καταναλωτού θα πρέπει να υπάρχει πλήρης αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων ή μειονεκτημάτων αυτών των τεχνολογιών. Ε, θα πρέπει να υπάρχει μια ε, διαφύλαξη των ε, στοιχείων του καταναλωτού, ταυτόχρονα με την προστασία των προσωπικών δεδομένων του καταναλωτού μαζί με την ανάγκη για την ε, προστασία του. Πιστεύουμε επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πάνελ, δεν υπάρχει ενημέρωση σε ε, ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν υπάρχει ένα σύστημα που επιτρέψει στους καταναλωτές να ανταποκρίνονται σε προβλήματα που ανοιχνεύουν στα προϊόντα τους και δεν υπάρχει ένας εναρμονμένος ορισμός σε σχέση με το τι καθιστά ελκυστικό προϊόν για τα παιδιά. Ευχαριστώ. Έχουμε φέρει και κάποια προϊόντα εδώ πέρα. Τα βρήκαμε στην ελληνική αγορά. Όλα σχολικά ήδη, ε, σχολικά ήδη πολλούνται. Αλλά μοιάζουν με παιχνίδια οπωσδήποτε. Είναι πολύ ελκυστικά για τα παιδιά. Το πρόβλημα είναι πως εάν δεν υπάρχει κοινός ευρωπαϊκός ορισμός του τι είναι ελκυστικό ένα ε, προϊόν για τα παιδιά θα είναι δύσκολο και για τις αρχές να κρίνουν το εάν αυτά τα προϊόντα εδώ πέρα μπορούν να διατεθούν στην αγορά και αν είναι ασφαλή ή όχι. Αυτό λοιπόν ζητάμε για κοινό ορισμό του ποια προϊόντα είναι ελκυστικά για τα παιδιά και κάποιες απαιτήσει ασφαλείας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, περνάμε τώρα αν έχουμε 10 δεύτερα να δείξω και την τελευταία διαφάνεια, τις δύο τελευταίες, όπως είπα, η γενική οδηγία ήταν επιτυχημένη, αύξησε τα επίπεδα προστασία των καταναλωτών, αλλά βεβαίως πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικοί οι κανόνες, χρειάζεται αποτελεσματικότερη υποπτία της αγοράς και βεβαίως πρέπει να δούμε και την ασφάλεια των υπηρεσιών. Ευχαριστώ και με συγχωρείτε. Τώρα δίνω τον λόγο στον τελευταίο ομιλητή. Η κυρία Edith Baxter, η οποία εκπροσωπεί την Business Europe και είναι και από τη Δανία, από ό,τι καλωσορίζω ιδιαίτερα. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, Κυρίε και κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ τους οργανωτές που προσκάλεσαν την Business Europe να παρουσιάσει τι απόψει τη στο εργαστήριο αυτό για την αναθεώρηση της Γενικής Οδηγίας για την Ασφάλεια των Προϊόντων. Και τα δύο αυτά ζητήματα ασχολούνται με το πώς θα έχουμε ασφαλή προϊόντα στην αγορά. Και δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία. Και η βιομηχανία αυτό θέλει. Εμείς θεωρούμε πως αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις, η βιομηχανία, οι πολίτες έχουν όλοι τα ίδια συμφέροντα. Μπορεί να μην ακολουθούμε τις ίδιες λύσεις, αλλά θα πρέπει να μπορούμε να επιτύχουμε τον στόχο. 1η Ιανουαρίου φέτος το λεγόμενο πακέτο των αγαθών ετέθη ενισχύ. Η Business Europe θεωρεί πως οι διατάξεις που υπάρχουν για την επιτήρηση της αγοράς και τον τηλεωνιακό έλεγχο θα οδηγήσουν σε πιο ασφαλή προϊόντα για τους πολίτες εάν τα κράτη-μέλη εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Όταν μιλάμε για ασφάλεια των προϊόντων, σημαντικό είναι να αντιληφθούμε πως υπάρχουν αρκετοί κρίκοι στην αλυσίδα και ο κάθε κρίκος έχει να παίξει τον ρόλο του. Το σύστημα βεβαίως είναι τόσο ισχυρό όσο ο κάθε κρίκος αυτής της αλυσίδας. Οπότε οι βουλευτές πρέπει να ασκήσουν πίεση στα κράτη-μέλη για να δώσουν επαρκείς πόρους για αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς και να φροντίσουν πώς θα ερμηνεύονται και θα εφαρμόζονται οι απαιτήσει με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις ε, χώρες. Οπότε, καλωσορίζουμε και τον ε, συντονισμό και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες από τις Βρυξέλλες όπως το είμαστε. Γεγονός είναι πως οι αυστηρότεροι κανόνες όπως παραδείγματος χάρη πιστοποίηση από τρίτους δεν σημαίνει αυτομάτως καλύτερα προϊόντα. Όλα, κάθε δοκιμή μπορεί να παραποιηθεί, κάθε πιστοποιητικό μπορεί να αντιγραφεί. Οι σοβαροί κατασκευαστές τι θα καταλήξουν να έχουν περισσότερο κόστος και γραφειοκρατία. Οπότε πρέπει οι αρχές να εξασφαλίσουν αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς και διασυνοριακή συνεργασία. Όμως, βεβαίως η εποπτεία δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Η βασική απέτηση είναι το προϊόν πρώτα απ' όλα να κληρώνει αυτά τα οποία λέει η νομοθεσία. Οπότε οι κανόνες πρέπει να είναι σαφείς και ξεκάθαροι η Business Europe καλωσορίζει την ευθυγράμμιση των οδηγιών προϊόντων με τις διατάξεις πλαίσιο που ορίζονται στο πακέτο των αγαθών. Η ευθυγράμμιση αυτή αφορά προϊόντα στον εναρμονισμένο τομέα. Οπότε χρειαζόμαστε αυτή την ευθυγράμμιση της Γενικής Οδηγίας για την Ασφάλεια των Προϊόντων με το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Κατά την άποψή μας δεν είναι τίποτα το επίγον. Αντιθέτως πιστεύουμε πως είναι το ζήτημα πρώτα απ' όλα η καλύτερη και ενιαία χρήση των υπαρχόντων εργαλείων. Επίσης, καλό θα ήταν πρώτα απ' όλα να έχουμε κάποια ευκαιρία με τις νέες απαιτήσει του πακέτου των αγαθών. Τι γίνεται στην πράξη. Εδώ πέρα σκεφτόμαστε ιδιαίτερα τις, επιχειρή... υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και την ίχνηλασιμότητα. Επιπλέον, η Γενική Οδηγία των Ασφάλων των Προϊόντων απαιτέλεσε έμπνευση και για τις διατάξεις επιτήρησης της αγοράς και για το πλαίσιο της απόφασης. Μάλιστα, τα πράγματα δεν ε, είναι τόσο άσχημα. Η Γενική Οδηγία λειτουργεί αρκετά καλά. Ο αριθμός των ειδοποιήσεων ΡΑΠΕΞ αυξάνεται. Αυτό οφείλεται στην ενημέρωση και στο ότι εστιαζόμαστε σε συγκεκριμένου τομεί, όπω παραδείγματο χάρη τα υφάσματα. Οπότε τα εργαλεία υπάρχουν. Όμω, λογικό είναι πάντα να σκεφτόμαστε το εάν η νομοθεσία που ισχύει λειτουργεί τελεία και αν μπορεί να βελτιωθεί η Κομισιόν. Κατέθεσε κάποιε προτάσει για τη βελτίωση τη Γενική Οδηγία και έχει υπάρξει δημόσια διαβούλευση online. Η Business Europe απάντησε στη διαβούλευση λίγο πολύ με αυτά τα οποία λέει και σήμερα. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται ένα συνεκτικό νομοθετικό πλαίσιο, οπότε σημαντικό είναι όταν έχουμε νέα νομοθεσία ή αλλάζει η φυστάμενη νομοθεσία να τις έχουμε σκεφτεί σοβαρά αυτές τις αλλαγές και να έχουμε αξιολόγηση αντικτύπου. Υπάρχουν άλλες οδηγίες που αφορούν διαφορετικές πτυχές ε, της σύνθεσης και σχεδιασμού των προϊόντων, όπως παραδείγματος χάρη αυτές που αφορούν τις χημικές ουσίες. Αυτές οι οδηγίες πρέπει να ληφθούν υπόψη έτσι ώστε οι απαιτήσει αυτές να εφαρμόζονται ενιαία διασυνοριακά. Εμείς θεωρούμε πως ένα συνολικό πολιτικό όραμα θα πρέπει να υπάρχει για την ομοθεσία προϊόντων, που ταυτόχρονα θα διασφαλίζει την ασφάλεια και το δημόσιο συμφέρον, καθώς και η ανταγωνιστική βιομηχανία. Χρειαζόμαστε ένα σταθερό νομοθετικό περιβάλλον με γνωστές απαιτήσει, αλλά θα πρέπει να μπορούμε να απαντήσουμε άμεσα σε κινδύνους που προκύπτουν. Επίσης, χρειαζόμαστε ευελιξία. Η καινοτομία είναι η λέξη κλειδί. Εάν έχουμε πολύ λεπτομερείς απαιτήσει, μπλοκάρουμε την καινοτομία. Η Business Europe θεωρεί πως σήμερα έχουμε ένα καλό μείγμα, δηλαδή η νέα προσέγγιση όπου περιέχονται οι απαραίτητες απαιτήσει συνδυάζεται με τη Γενική Οδηγία που είναι ένα δίκτυο ασφαλείας για τα μη εναρμοσμένα προϊόντα στην περίπτωση που έχουμε κινδύνους οι οποίοι είναι άγνωστοι ή είδαν απρόβλεπτοι. Επιπλέον, η Γενική Οδηγία αποτελεί μια ομπρέλα για το επίπεδο ασφάλειας προϊόντων μη εναρμονισμένων. Η χρήση προδιαγραφών βοηθάει και τους κατασκευαστές να επιτύχουν το απαιτούμενο ποσοστό ασφαλείας και τις συγκεκριμένες απαιτήσεις. Στην πράξη, τα, οι είναι και θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι εθελοντικές. Η Κομισιόν πρότεινε να υπάρχει ένας πιο γρήγορος τρόπος διατύπωσης εντολής για τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές σε σχέση με τη Γενική Οδηγία και να μπορούν να οριστούν έτσι πιο συγκεκριμένες απαιτήσεις. Βεβαίω, το να οριστεί η εντολή δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει γρήγορα. Πρέπει να υπάρξει πρώτα απ' όλα διαβούλευση με του ενδιαφερομένους και βεβαίω δεν θα πρέπει η εντολή αυτή να πάει σε λεπτομερείς και σχεδόν υποχρεωτικές απαιτήσει. Εάν και όταν έχουμε μόνιμες τέτοιες απαιτήσει, θεωρούμε πως θα πρέπει να ακολουθεί η κανονική νομοθετική διαδικασία καθώς η επιτροπολογία μπορεί να μην είναι τόσο δημοκρατική διαδικασία όταν χρειάζεται να ασχοληθεί με κάτι περισσότερο από τεχνικέ λεπτομέρειε. Όσον αφορά την πιθανή ευθυγράμμιση με τι υποχρεώσει των επιχειρήσεων, εμεί είμαστε υπέρ τη αναλογικότητα. Χρειαζόμαστε ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο εάν είναι να καλύψουμε όλα τα προϊόντα και όταν μιλάμε για εχνηλασιμότητα και οι διανομής έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν. Πρέπει να ξέρουν πού αγόρασαν ένα προϊόν και να δώσουν αυτή τη πληροφορία στις αρχές όταν τους το ζητάνε. Οπότε είναι και ζήτημα του να οριστούν οι υποχρεώσεις των διαφορετικών επιχειρήσεων χωρίς να αντιγράφουμε κατά λέξη την απόφαση πλαίσιο του πακέτου των αγαθών. Συμπερασματικά λοιπόν είμαστε υπέρ της αποτελεσματικής και ενιαίας επιτήρησης αγοράς ενός σταθερού νομοθετικού πλαισίου. Δεν χρειάζεται άμεση αναθεώρηση της γενικής οδηγίας εάν είναι σύμφωνη με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, ευελιξία και αναλογικότητα, λέξεις κλειδιά και για μόνιμε απαιτήσει προϊόντων εμεί προτιμούμε δημοκρατική και διάφανη διαδικασία. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ όλου σα. Ζητώ συγγνώμη γιατί σα πίεσα πολύ για τη βιασύνη. Έχουμε κανένα δύο λεπτά ακόμα διότι στι 12.30 και είναι άλλη συνεδρίαση. Κάποιος συνάδελφο θέλει να πάρει το λόγο. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μάρκ Ταραμπέλα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν ξέρω το ερώτημά μου απευθύνεται προς τον κύριο Τεκούνιγκ ή στον κύριο Σόρο της Γενικής Διευθύνσης ΣΑΜΚΟ όσον αφορά την, το Rapid Exchange, τη διαδικασία αυτή. Δηλαδή μπορούν τα κάτι μελη να ζητήσουν πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ενημερώσουν τα κάτι μελη όταν υπάρχει από προϊόν που, που απειλεί την υγεία. Θα ήθελα να ξέρω αν τα κάτι μελη χρησιμοποίησαν τη διαδικασία. Εάν ναι, ε, συμβαίνει συχνά και σε περίπτωση που ε, κινητοποιείται το, σύστημα υπάρχει αντίδραση από τα άλλα κράτη-μέλη. Όταν διαπιστώνεται ότι υπάρχει κίνδυνος για την υγεία ε, μπορεί να στείλει εντολή στο κράτη-μέλη να τα υποχρεώσει να αποσύρουν ε, το προϊόν από την αγορά ή τα κράτη-μέλη έχουν δυνατότητα να αντιδράσουν ανάλογα με τη βούλησή τους όπως θεωρούν ότι πρέπει. Καλώς. συντομία, έμαθα ότι από ε, τον Ιανουάριο αυτού του έτους δεν ε, μεταφράζονται οι ανακοινώσει της ΡΑΠΕΞ. Και θα ήθελα να μου πείτε τι πιστεύει η Κομισιόν γι' αυτό. Γιατί φαίνεται ότι σε μια κρόση δεν δόθηκε, σε κάποια αίτηση, συγγνώμη, δεν δόθηκε κάποια απάντηση. 15 seconds. Έχετε 15 δευτερόλεπτα να Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους της κυρίας Κορχόλα, έχω ένα ερώτημα. Αφορά τα προϊόντα που αγοράζονται με τον υπολογιστή online. Έχουμε ανησυχίες και θεωρούμε ότι η υποπτή αυτών των προϊόντων δεν είναι πολύ καλή. Μπορεί να επιληθεί το πρόβλημα αυτό των προϊόντων που αγοράζονται online. Ποιε είναι οι νομικές στοιχείες τη εποπτεία των προϊόντων που αγοράζονται online. Να κάνουμε το εξή. Δεν έχουμε χρόνο για τις απαντήσεις. Θα έρθω σε επαφή με τους υπευθύνου που ξέρουν τις απαντήσεις. Θα σα δώσω τις απαντήσεις αργότερα. Και οι Σκιώδης και εγώ θα εξακολουθήσουμε το διάλογο επί των σημαντικότατων αυτών ζητημάτων. Ευχαριστώ όλους που ήρθαν. Ζητώ συγγνώμη για την χρονική πίεση και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Σας εύχομαι καλή σας μέρα. Γεια σας.